Uh, ladies and um, Κυρίες και κύριοι, μόνο η σκιώδεις και ο εισηγητής είναι εδώ, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Να σας ζητήσω να καθίσετε. Σας καλωσορίζω. Κάποιες σύντομες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ξέρετε ότι όπως συμβαίνει πολύ συχνά στις συνεδριάσεις μας α, ε, ε, αναμεταδίδεται η συνεδρίαση αυτή στο διαδίκτυο. Έγινε μια συνάντηση στην Κρακοβία, ξέρετε, όπου είχαμε μια ισχυρή παρουσία. Ήμασταν συνδιοργανωτές και αυτό ε, αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο και αυτό έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσουν οι πολίτες τις προτεραιότητες που έχουμε για την εσωτερική αγορά. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι αυτό το φόρουμ για την ενιαία αγορά ήταν μεγάλη επιτυχία. Υπήρξε πολύ δραστήρια συμμετοχή, 80 μέλη του Κοινοβουλίου, πολλά μέλη της δικής μας Επιτροπής εισηγητές, πρόεδροι ομάδας εργασίας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την πρακτική. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια νέα δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την προσπάθεια την οποία κάναμε μέχρι τώρα. Περιλαμβάνεται στην πρώτη σελίδα του newsletter το οποίο εμείς συντάσσουμε. Ελπίζω συνιστώ να το διαβάσετε. Όπως είπα και χθες, σήμερα θα συζητήσουμε τέσσερις από τις 20 βασικές ανησυχίες των πολιτών. Το, το roaming, τα ψευδεπίγραφα προϊόντα, τους βασικούς λογαριασμούς πιστοτικούς στις τράπεζες, Ελπίζω λοιπόν αυτό να δείχνει ότι προσπαθούμε με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Έχουμε επίσης και τη σύνοψη των ε, ομάδων εργασίας της Κρακοβίας, της συνάντησης του Φόρουμ στην Κρακοβία δηλαδή, και κάποια πρώτα συμπεράσματα που δεχθήκαμε και ζητάμε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε γρήγορη εφαρμογή της ενίας πράξης. Ξέρω ότι η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί με το αίτημα αυτό. Ξέρω ότι η κυρία Μέρκελ είναι σήμερα εδώ και γι' αυτό κάποιοι συνάδελφοι που ίσως τη συναντήσουν μετά να επιμείνουν προς την κατεύθυνση αυτή απέναντί της. Λοιπόν, η ημερήσια διάταξη τώρα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις δεκτή. Έχουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11ης Ιουλίου στους φακέλους σας. Σχόλια τα οποία έχετε παρακαλώ να τα στείλετε μέχρι αύριο το μεσημέρι στη γραμματεία, αλλιώς θα θεωρηθούν δεκτά. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη τη σημερινή. Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 11. Θα αντικατασταθώ όμως γιατί πρέπει να, να συναντηθώ με τον Βρετανό Υπουργό Εμπορίου που θα είναι στις Βρυξέλλες. Με μεγάλη χαρά γιατί ξεκινάμε τη συζήτηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής As I think you will all know, we did a a very full strategic report on that under the leadership of Edvard Kozisnik. I'm pleased to. Τα θέματα της τυποποίησης προκαλούν ενδιαφέρον. Προετοιμάζεται η νομική πρόταση η οποία θα συνταχθεί από την κυρία Κόμη Όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς κάνουμε μια στρατηγική προσπάθεια, συνεργάζεται και ο κ. Κρόιτσμαν και άλλοι συνάδελφοι. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει καταρχάς την αξιολόγηση των συνεπειών εφαρμογής της πρότασης. Θα δώσω το λόγο στις κυρίες, κυρίες Μπρίνκμαν και Βάισερ Χόρνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ζητήσω επίσης και από την κυρία Κόμη να κάνει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις αν θεωρεί είναι η πρώτη δυνατότητα που έχει για να μιλήσει στην Επιτροπή. Λάρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Κόμη, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αναθεωρήσεων την οποία προτείνει για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ξεκινάμε την διακοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός νέου κανονισμού για την τυποποίηση στην Ευρώπη. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει όπως είπε ο Πρόεδρος εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο με την επεξεργασία της έκθεσης πρωτοβουλίας όπως βλέπετε και οι σκιώδεις εισηγητές είναι οι ίδιοι, απλά έχουμε αναλάβει διαφορετικούς ρόλους με αυτούς που είχαμε στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα παρουσιάσει το έγγραφό της λεπτομερώς, έλαβε υπόψη πολλές από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό για μας είναι ένας επιπλέον λόγος ευχαρίστησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει όλο και περισσότερο το ρόλο του ως συνομοθέτης και ακριβώς ε, μπορεί να ε, προτείνει και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις επιθυμίες και να καταγράψει τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Η εσωτερική αγορά πρέπει να απαλλαγεί από τα εμπόδια που την ε, παρεμποδίζουν ακριβώς και νομίζω ότι μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα τυποποιήσεις θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των δυσκολιών των οικονομικών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Η γενική όρια αναφοράς δεν είναι μια ανακύκλωση αν θέλετε του πακέτου και του συστήματος αλλά κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις. Εγώ στα πλαίσια αυτής της ευκαιρίας δεν θα ήθελα να κάνω κάποιες τελικές προτάσεις και κάποιες επακριβήσεις να δώσω κατευθύνσεις. Πρώτα θα ήθελα να σας ακούσω, πρώτα θα ήθελα να ακούσω τους διάφορους εμπλεκομένους και μετά θα σας κάνω την πρόταση ψηφίσματος. Την 23η Νοεμβρίου, στα πλαίσια της ακροάσεως την οποία θα οργανώσουμε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συλλέξουμε τις διαφορετικές απόψεις και να αναπτύξουμε νέες προτάσεις. Θα περιοριστώ στο να συμμεριστώ μαζί σας μια πρώτη αντίδραση στο πακέτο αναθεωρήσεων υπογραμμίζοντας τα βασικά θέματα στα οποία θα σταθούμε τους επόμενους μήνες. Όπως είχα ήδη τη δυνατότητα να πω επανειλημμένα στο παρελθόν και όπως πιστεύουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της προτάσεως ε, θα πρέπει να διατηρηθούν και ακριβώς το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ιδιωτικός χαρακτήρας του συστήματος, σαν παράδειγμα. Ο εθελοντικός χαρακτήρας, όπως επίσης και το θέμα της εθνικής αντιπροσωπείας. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να εμείνουμε. Νομίζω ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι καταρχάς ιδιωτικό και η ανάπτυξη των, των στάνταρ των ε, επιπέδων τυποποίησης θα είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να αποδεικνύεται άμεσα σε εθνικό επίπεδο. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω μία κάποια αμφιβολία γιατί πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να κρυθούν με τον ίδιο τρόπο. Ή έχουμε να κάνουμε με ασθενείς ε, εμπλεκόμενους στο σύστημα, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να παρέμβει στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, προστατεύοντας ακριβώς τα κοινωνικά συμφέροντα και εξυπηρετώντας συγκεκριμένη περίπτωση της μικρομεσαίας. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια σωστή διαβούλευση γιατί η πρόθεσή μας και στην οδηγία και στον κανονισμό ε, είναι να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο. Θεωρώ ότι η αντιπροσώπευση των μικρομεσαίων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα έλεγα είναι το υπόστρωμα αλλά και το σύνολο ουσιαστικά της δομής της ευρωπαϊκής οικονομίας και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν καλύτερα. Θα δώσω το λόγο τώρα πάλι στον Πρόεδρο, θα αφήσω το λόγο στον Πρόεδρο και μετά στην Επιτροπή για να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καμή. Θα σας ξαναδώσω το λόγο αργότερα για να μας πείτε τα σχέδιά σας για την ακρόαση και το χρονοδιάγραμμα για την έκθεσή σας. Όμως σήμερα το πρωί τώρα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπρίγμα νομίζω θα ξεκινήσει. Φαντάζομαι ότι έχετε αντίγραφο των διαφανειών της. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Κάμη, για την πρώτη παρουσίασή της όσον αφορά την άποψη του Κοινοβουλίου για το πακέτο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμεριζόμαστε την άποψή της για τη σημασία που έχει να χτίσουμε πάνω στο υπάρχον σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης και να μην αλλάξουμε ριζικά το σύστημα όπως ε, ήταν αρχικά η πρόταση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω τώρα να σας παρουσιάσω την ε, έκθεση αντικτύπου η οποία έγινε και αποτελεί ένα νομικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το πακέτο έτσι όπως εγκρίθηκε την 1η Ιουνίου του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή α είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα κύρια στοιχεία της διαβούλευσης αυτής όπως επίσης και ο διάλογος με τους ειδικού είναι πράγματα τα οποία βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αυτή. Έχετε πρώτα απ' όλα τη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα Μάρτιο με Μάιο 2010 για να ετοιμαστεί η έκθεση αντικτύπου. Στη συνέχεια είχαμε τη λευκή ε, βίβλο για τον εξυγχρονισμό της ηλεκτρονικής ε, τυποποίησης το 2009. Στη συνέχεια είχαμε το Express Report το 2010 από ειδικού και μετά είχαμε και την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και διάφορα συμπεράσματα του Συμβουλίου ιδιαίτερα του Φεβρουαρίου του 2011, όπου αναφέρεται ότι η διαδικασία τυποποίησης πρέπει να επιταχυνθεί, να απλοποιηθεί και να γίνει πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία να προσαρμόζεται η τυποποίηση στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα και στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στο περιβάλλον. Όλες αυτές οι απόψεις των ειδικών και μη μας κάνουν να συμπεραίνουμε ότι η χρήση της ευρωπαϊκής τυποποίησης ως μέσο για την εκπόνηση πολιτικής αποτελεί μια επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που χρησιμοποιείται στην εσωτερική αγορά, για την διαλειτουργικότητα. Όμως η δημόσια διαβούλευση και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντοπίζει ορισμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ακόμα. Στην έκθεση αντικτύπου έχουμε εντοπίσει τρία κυρίως προβλήματα, τα οποία αντικατοπτρίζονται ε, στη συνέχεια στο νομικό μέσο. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία έγκρισης ε, των ευρωπαϊκών ε, τύπων δεν προχωράει αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην ε, εκπόνηση της τυποποίησης αυτή στην Ευρώπη. Και το τρίτο είναι ότι διάφορα φόρα και κονσόρτια και οι δικές τους προδιαγραφές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις. Όπως συμβαίνει συνήθως, την έκθεση αντικτύπου, έχοντας εντοπίσει τα κύρια προβλήματα, εξετάσουμε στη συνέχεια τι επιλογές έχουμε για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαδικασία έγκρισης της ευρωπαϊκής τυποποίησης, επειδή πηγαίνει ενεργά, έχουμε τρεις επιλογές. Για την πρώτη θα έπρεπε πρώτα να σας πω ότι υπάρχουν τέσσερα στάδια στην διαδικασία έγκρισης ε, τυποποίησης. Το πρώτο είναι η προετοιμασία της εντολής και η θετική άποψη της Επιτροπής μέσω μιας οδηγίας του 2004, κάτι το οποίο παίρνει 6 με 12 μήνες. Το δεύτερο στάδιο είναι η αποδοχή της εντολής από την Οργάνωση Ευρωπαϊκής Τυποποίησης και έτσι αρχίζει και η δουλειά. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αξιολογή. Μετά από τρεις μήνες ε, κατά μέσο όρο, πάει από τρεις μάλλον μέχρι 13 μήνες περίπου. Έπειτα προχωράμε στην τυποποίηση αυτή ή καθεαυτή και μετά χρειάζονται και δύο ακόμα χρόνια για να καταλήξουμε. Το τελευταίο, το τέταρτο στάδιο είναι η αποδοχή της τυποποίησης και ενσωμάτωσή της στην ε, διαδικασία. Μπορούμε να συνοψίσουμε ότι η όλη διαδικασία από τη στιγμή της εντολής παίρνει κάλλιστα τρία χρόνια και μερικές φορές και πολύ περισσότερο. Εξετάσαμε λοιπόν τρεις επιλογές για να μειωθεί το χρονικό αυτό διάστημα το οποίο χρειάζεται η διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης από τη στιγμή που λαμβάνει έτοιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη επιλογή, ένα α, είναι να βάζουμε προθεσμίες για ε, την τυποποίηση αυτή. Να βάζουμε ε, προθεσμίες για την εντολή. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, να αναπτύξουμε πιο γρήγορα την τυποποίηση, η ανταγωνιστικότητα θα ενισχυθεί έτσι και οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν και κόστος. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στον... Ε, ε, στο, ότι δεν θα υπάρχει κατακαιρματισμός στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν πιο γρήγορα να, αναπτύσσονται, να αναπτύσσεται η τυποποίηση αυτή, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες βέβαια. Μέρος τώρα της επιλογής αυτής θα ήταν και η εισαγωγή οικονομικών κινήτρων για να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας, δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα να στραφεί περισσότερο σε ένα σύστημα καλύτερων επιδείσεων ε, βασιζόμενοι σε δείκτες και στην απλοποίηση. Η άλλη εναλλακτική λύση, ένα β, είναι να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα standards. Έτσι η υπηρεσία αυτή θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και θα μπορούσε να δράσει και σαν γραμματεία για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Κοιτώντας διαφορετικά την αρχή για την εθνική εκπροσώπηση. Όμως είναι σαφές ότι μια τέτοια υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη στήριξη των εθνικών σωμάτων τυποποίησης. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει συνένεση, θα είναι ακόμα αναγκαία και σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον με την επιλογή αυτή θα έχουμε επιπλέον κόστος στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και τέλος θα υπάρχει και αρνητικός αντίκτυπος στο κόστος ενώ θα υπάρχει θετικός αντίκτυπος στην ποιότητα της διαδικασίας τυποποίησης. Αν και αυτό αμφισβητείται κάπως, γιατί είναι ένα ζήτημα οι δραστηριότητες τυποποίησης, όπου ο κύριος φορέας είναι ιδιωτικό θα μπορούσε να χρηματοδοτείται από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, δεδομένου ότι η σημερινή δομή ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές ανάγκες. Υπάρχει και η τρίτη εναλλακτική λύση και αυτή είναι η εισαγωγή διαδικασιών απλοποιημένων που διέπονται από διαφάνεια για ό,τι στάνταρτ ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει πιστεύουμε ένας θετικός αντίκτυπος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης θα μπορεί έτσι να προλαμβάνει τις ε, αιτήσει που θα έρχονται και θα υπάρχει μια πιο σύντομη περίοδος αποδοχής των αιτήσεων αυτών. Πιστεύουμε ότι γενικά θα υπάρχει θετικός αντίκτυπος χωρίς να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την ε, εναλλακτική αυτή λύση. Το μόνο αρνητικό μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι θα εφαρμόζεται μόνο σε εναρμονισμένες ε, προδιαγραφές ενώ δεν θα επηρεαστεί καθόλου ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουμε στην υπόλοιπη τυποποίηση. Συνεπώς, η προτιμότερη λύση για μας, μετά την ανάλυση μας, είναι η 1α και η 1γ. Εξετάζουμε τώρα το δεύτερο πρόβλημα, που είναι η μη ικανοποιητική εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μη επαρκής. Εδώ εξετάζουμε ναι, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από πλευρά τη κοινωνία. Και εδώ πάλι έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι η 2α, που είναι να διευκολύνουμε την άμεση εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης απαιτεί να κατανοεί κανείς καλά την τεχνική πτυχή της τυποποίησης. Μια συνεχιζόμενη συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις απαιτεί πολύ μεγάλη δέσμευση και από πλευράς χρόνου που θα πρέπει να διαθέσουν οι ενδιαφερόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έπειτα η εκπροσώπηση αυτή άμεση είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να μπορεί να επηρεάζει πολύ συγκεκριμένα την εκπόνηση της τυποποίησης. Οι τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας όμως που είναι πολλές έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δύσκολη άμεση αυτή η εκπροσώπηση. Έπειτα σε γενικότερο επίπεδο η εξατομικευμένη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην διανέμεται αποτελεσματικά η πληροφόρηση σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αυτές δηλαδή που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία τυποποίησης. Και τέλος η επιλογή αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί πολύ ο αριθμός των συμμετοχόντων στη διαδικασία τυποποίησης Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος τελικά στην ταχύτητα με την οποία θα προχωράει η διαδικασία τυποποίησης. Οπότε, δεν διακόπτει η ομιλήτρια. Προχωράμε στην επόμενη λύση, 2β, που ε, δίνει το δικαίωμα ψήφου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους ώστε να εκπροσωπούνται με την ψήφο τους στις οργανώσεις. Το δικαίωμα αυτό ψήφου σε οργανώσεις όμως εκτός των εθνικών ε, υπηρεσιών τυποποίησης είναι κάτι που πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθεί και να εγκριθεί με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η εναλλακτική λύση δεν είναι και πολύ εφικτή. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη εναλλακτική 2Γ, που είναι να ενισχύσουμε την ε, ε, θέση εκπροσώπησης διαφόρων ε, οργανισμών μέσω ενός δικαιώματος λειτουργίας. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε οργανώσεις που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους. Έτσι ενισχύεται ο ρόλος τους στην διαδικασία τυποποίησης. Για να λύσουμε λοιπόν το δεύτερο πρόβλημα, έχουμε επιλέξει την λύση 2Γ. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο πρόβλημα, που είναι η συμμετοχή στις ε, δημόσιες συμβάσεις και εδώ πάλι έχουμε τρεις λύσεις. Η μία είναι να ξαναδούμε την απόφαση 87-95 όσον αφορά την τυποποίηση σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και πιστεύουμε ότι αυτή η λύση δεν συνοδεύεται από νομική βεβαιότητα και δεν στηρίχτηκε κατά την διαδικασία διαβούλευσης. Η δεύτερη λύση, 3β, θα ήταν να επιτρέπουμε referencing σε δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή να μπορούν να επιλέγονται κάποια κονσόρτια και κάποια φόρα βάσει μιας δίκαιας νομικής βάσης. Αυτό όμως θα οδηγήσει στην τάση κατακαιρματισμού της αγοράς. Και δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει τελικά την εσωτερική αγορά. Ελοχεύουν εδώ κάποιοι κίνδυνοι, οπότε η λύση αυτή 3Β μάλλον θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ερχόμαστε τώρα στην εναλλακτική 3Γ που είναι σε συγκεκριμένα κοσόρτια να δώσουμε το καθεστώς του αναγνωρισμένου σώματος τυποποίησης. Αυτή η αναλλακτική λύση βέβαια απαιτεί πολύ καλό έλεγχο για να έχουμε εγγυήσει όσον αφορά τα φόρα και τα κοσόρτια αυτά. Τελικά, η λύση αυτή δεν επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Συμπέρασμα για το τρίτο πρόβλημα, η προτίμησή μας πηγαίνει στη λύση 3β. Ερχόμαστε τώρα στα άλλα στοιχεία που εξετάσαμε κατά την μελέτη μας αντικτύπου. Η δυνατότητα απλοποίησης και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει. Πιστεύουμε ότι ένα απλοποιημένο νομικό πλαίσιο θα βοηθούσε περισσότερο. Και γι' αυτό σήμερα ερχόμαστε με μια ε, νέα πρόταση απλοποιημένου ενιαίου πλαισίου αντί για τα τρία που είχαμε πριν. Εδώ στη διαφάνεια αυτή βλέπετε διάφορα θέματα. Αλλά από αυτά θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στο τελευταίο, δηλαδή την ευρωπαϊκή τυποποίηση όσον αφορά τις υπηρεσίες. Η οδηγία για την κοινοποίηση έχει να κάνει μόνο με την τυποποίηση προϊόντων. Και υπάρχουν επιτροπές εκπροσώπων κρατών μελών που λένε ότι με την οδηγία αυτή δεν μπορούν να προτείνουν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητάει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης να ε, φτιάχνει τυποποίηση για τις υπηρεσίες. Εδώ πιστεύουμε ότι χρειάζεται ευθυγραμμισμός και απλοποίηση των διαδικασιών για όλες τις εντολές που φτάνουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης ανεξάρτητα από το θέμα και συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητα να ζητάνε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης να εκπονεί τυποποίηση και για τις υπηρεσίες στο νομικό κείμενο. Η δημόσια διαβούλευση έδειξε ότι η δυνατότητα αυτή στηρίζεται πάρα πολύ. Η μελέτη αντικτύπου στο παράρτημα 5 συμπεριλαμβάνει και κάποιες άλλες επιλογές που δεν έχουμε επιλέξει, δεν χρειάζεται να σας τις αναφέρω, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά όλες αυτές ε, οι επιλογές που απορρίφθηκαν υπάρχουν στη διαφάνεια αυτή και εξηγούνται στο παράρτημα 5. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την μελέτη αντικτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για κανονισμό προκειμένου να αντικατασταθεί οι διάφορες αποφάσεις ε, της Επιτροπής και η οδηγία μέρος της οδηγίας μάλλον 9834 ναι, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αλλάζει καθόλου έτσι δεν επηρεάζεται από την πρόταση αυτή και έχουμε επίσης προτείνει και τροποποίηση διαφόρων τομεακών οδεϊγιών σχετικά με την εναρμονισμένη τυποποίηση. Η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει τα κύρια στοιχεία του νέου κανονισμού που προτείνουμε. Θα επεκτείνουμε τους ορισμούς και το εύρος που καλύπτει ο κανονισμός και στις υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε λοιπόν να δώσει εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης προκειμένου να ετοιμάσει τυποποίηση για στήριξη και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Στη συνέχεια έχουμε δύο άρθρα για την συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Αυτό δεν αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα νομικά μέσα που είχαμε στο άρθρο 5 θέλουμε να αναφέρουμε τη σημασία που έχει η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Και επίσης αναφέρουμε και ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή η τι οργανώσεων πρόκειται με κριτήρια τα οποία καλύπτει το παράρτημα 3 του κανονισμού. Ο κανονισμός επίσης προβλέπει περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, όπως επιπλέον και μεγαλύτερη προβολή των προτεραιοτήτων που υπάρχουν στην τυποποίηση μέσω προγραμμάτων που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα ένα κατάλογο μελλοντικών εντολών. Εδώ δουλεύουμε πάνω στην πρώτη εκδοχή αυτού του προγράμματος και πιστεύουμε ότι στα τέλη της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο μια ανακοίνωση σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τη σημαντική τυποποίηση που έχει ζητηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή του χρόνου. Το άρθρο 7 έχει να κάνει με έτοιμα στο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και υπάρχουν προτάσεις για το πώς θα μειωθεί η διοικητική διαδικασία. Άρθρο 7. Το άρθρο 8 αναφέρεται στις ενστάσεις όσον αφορά την εναρμόνιση. Είναι μια διαδικασία η οποία θα χρησιμοποιείται εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο, όπως λέει το άρθρο 22. Στη συνέχεια, το σημαντικό Και το στοιχείο καινοτομία του κανονισμού είναι η δυνατότητα αναγνώρισης προδιαγραφών ICT για δημόσιες συμβάσεις. Αυτά αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10. Ακούμε τις προτάσεις όλων των χωρών μελών και άλλων ενδιαφερομένων. Υπάρχει μια πλατφόρμα που θα γνωμοδοτεί προετοιμάζεται αυτή την εποχή. Πρόκειται για μια ευρεία πλατφόρμα όπου βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ποιοι θα συμμετέχουν. Ποιοι θα κληθούν ως μέλη στην πλατφόρμα αυτή. Του χρόνου θα αρχίσει ήδη να λειτουργεί και θα έχει έναν πολύ σημαντικό γνωμοδοτικό ρόλο να παίξει όσον αφορά την Επιτροπή, θα την γνωμοδοτεί δηλαδή. Υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό παράρτημα 2 που αναφέρει τα κριτήρια ποιότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να αναγνωρίζεται η τυποποίηση ICT όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές είναι οι βασικές αρχές και αναφέρεται μεταξύ άλλων η σχέση της τυποποίησης με τα δικαιώματα διανοτικής ιδιοκτησίας. Η επόμενη διαφάνεια αναφέρεται στη χρηματοδότηση. Υπάρχουν τα άρθρα 11 έως 13, τα οποία περιλαμβάνουν τη γενική βάση για τις δραστηριότητες που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης. Με τη, σε τη βάση, με τι ποσά καταποκοπή κλπ. Αναφέρεται και η χρηματοδότηση βέβαια ευρωπαϊκών οργανισμών που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους όσον αφορά τις δραστηριότητε τους. Αυτά αναφέρονται στα άρθρα που σας είπα, που είναι και στη διαφάνεια. Ο κανονισμός επίσης περιλαμβάνει και τους κανόνες επιτροπολογίας για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Πρόκειται για τα άρθρα 16 και 17. Όπως επίσης και το ρόλο μιας νέας επιτροπής που ο κύριος ρόλος της θα είναι να ασχολείται με τις ενστάσεις όσον αφορά την εναρμόνιση της τυποποίησης. Θα γνωμοδοτεί, θα συμβουλεύει όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας, για παράδειγμα. Και έτσι φτάνω στο τέλος της παρουσίασής μου, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην εξέταση των προτάσεών μας αυτών. Ελπίζουμε πραγματικά ότι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα καταλήξουν σε συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες. Για μας το ιδανικό θα ήταν να έχει εγκριθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Η πρόταση αυτή, καταλαβαίνετε, ότι δεν πρέπει να τη δούμε μόνο στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ευρώπη το 2020, αλλά είναι και θέμα ενιαίας πράξης για την ενιαία αγορά δηλαδή. Πρόκειται για τα 12 θέματα που αναφέρονται εκεί και που πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε επικοδομητική συνεργασία για ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Well, thank you very much indeed. Um, Εγώ ευχαριστώ. Όντως στην παρουσίασή σας παρουσιάζεται το τι θα πρέπει να κάνει η αξιολόγηση επιπτώσεων, να δίνει δηλαδή τις επιλογές για τις πολιτικές που προτείνετε. Αναλύσατε και ποιες είναι οι αδυναμίες, αλλά και ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της πρότασης. Συνάδελφοι, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την αξιολόγηση αυτή, για να ξεκινήσει κιόλα. Αλλά νομίζω ότι τελικά ε, έχουμε μόνο χρόνο για ένα γύρο σχολείων. Βεβαίως, αν θεωρείτε ότι κάτι έχει παρελθεί, Ευχαρίστω να το ακούσουμε, αλλά στι λεπτομέρειε θα μπούμε άλλη στιγμή. Να καλωσορίσω και δύο ε, ομάδε επισκεπτών από την κυρία Βάιλερ. Έχουμε ε, από τον Νόεχοφ, από το Συμβούλιο του ΚΕΝΕΣ, μια ομάδα ε, επισκεπτών και μια ομάδα επιχειρηματιών από το Κάσελ. Ε, νομίζω ότι είναι χρήσιμε οι συζητήσει που ακούτε σήμερα, γιατί όλα αυτά που γίνονται μπορούν όντω να επηρεάσουν και τι δικέ σα εταιρείε. Αυτό τώρα που θέλω να κάνουμε είναι να δώσουμε το λόγο στους σκιώδε. Η κυρία Καμία έκανε τα... Λαμία έκανε τα βασικά τη σχόλια, οπότε ο κύριος Κρόιτσμαν θέλει το λόγο. Α, κάποιοι δεν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε λοιπόν λίγα λόγια από τους σκιώδες και μετά θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια για μια τελευταία κουβέντα. Η κυρία Σαλντεμόσα. Θα μιλήσω στα δανέζικα, πρόεδρε, αν μπορώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εξαιρετική πρόταση που υπέβαλε. Όντως έχει λάβει υπόψη πολλά στοιχεία που είχαμε παρουσιάσει και εμείς στην έκθεση της Επιτροπής μας. Οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Η κυρία, α, κυρία Κόμη πρέπει να πω ότι πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο στην, για τη λεπτομέρεια του πράγματος για να δούμε αν μπορούμε τελικά να βελτιώσουμε σε κάποια σημεία την πρόταση της Κομισιόν. α ας, ας δούμε κάποια πράγματα για τις προτεραιότητες των σοσιαλιστών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία τυποποίησης και η οργάνωσή τη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το δημόσιο συμφέρον σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να δούμε πιο στενά το πώ διατυπώνεται όλο αυτό. Στην πρόταση λέει ότι θα πρέπει να δούμε την εκπροσώπηση προφανώ από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, ενδιαφερόμενους φορείς από την κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο στενά, να το ορίσουμε καλύτερα. Και θα μπορούσαμε ίσω να κάνουμε και πιο συγκεκριμένε προτάσει σε ό,τι αφορά τι οργανώσει, όχι μόνο των καταναλωτών, ε, των ε, εργαζομένων, α πούμε. Και αυτοί θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και τέλο, ό,τι αφορά την ε, ταχύτητα. Πολύ συχνά συζητούμε το γεγονό ότι αυτή η διαδικασία τυποποίηση είναι λίγο αργή. Και νομίζω ότι η Κομισιόν το έλαβε αυτό υπόψη της στην πρότασή της. Πάρα όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την εργασία αυτή και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο οικονομικά. Θα πρέπει ίσως να καταστήσουμε δυνατή την ε, ύπαρξη βοήθειας ό,τι αφορά την ε, ερμηνεία. Όχι μόνο, να μην μιλούμε δηλαδή μόνο με οικονομικούς όρους, ε, είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ε, καλή εποπτεία όλες αυτές τις ε, διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε εγώ πραγματικά αναμένω, προσβλέπω στην συνεργασία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε τελικά σε ένα καλό νομοθετικό κομμάτι πλαίσιο για αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρότσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, η σημασία των προτύπων για την εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική, δεν χρειάζεται να την τονίσω εγώ. Τα κοινά πρότυπα βοηθούν την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι προσπάθειε μπορούμε για να βελτιώσουμε το, το... το... τη διαδικασία αυτή και να μπορέσουμε να καλύψουμε τα ε, συμφέροντα και τι ανάγκε όλων. Βεβαίω, τα πράγματα έχουν αλλάξει όλο και, λιγότερα έντυπα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται, μια που, μια που τεχνολογίες, ε, ε, η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς. Ε, οπότε η διαδικασία στο μέλλον θα πρέπει, της τυποποίησης θα πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορη. Ε, βεβαίως αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει την ποιότητα. Γι' αυτό υπάρχει, έτσι πρέπει να δούμε με κάποια, κάποιο σκεπτικισμό το θέμα των προθεσμιών. Τώρα, η, αυτό που προτείνεται στην πρόταση είναι νομίζω αρκετά σκόπιμο. Ε, θα πρέπει ίσω να περιοριστούν κάποια πράγματα εφόσον υπάρχει ανάγκη και εφόσον αυτό είναι δυνατό. Τώρα, για, την, για τον ορισμό των προϊόντων, ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό με αναλογία ένα προ ένα μεταφορά στι αντίστοιχε ε, υπηρεσίε. Βεβαίω ε, θα πρέπει να δούμε τι ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χαίρομαι που η Κομισιόν στην πρότασή τη έχει συμπεριλάβει περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην διαδικασία της τυποποίησης, γιατί τώρα ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συνήθως ε, δεν επωφελούνται από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, περισσότερο. Η συμπερίληψη λοιπόν των επιχειρήσεων και σε εθνικά βήματα, καθώς επίσης και οι ε, ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, νομίζω ότι έχουν ε, ρόλο να παίξουν σε αυτή τη διαδικασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, να υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες συμμετοχής και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως γίνεται με, τις ε, με τους μεγαλύτερους οργανισμούς ο στόχος θα πρέπει να είναι να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση, συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Γενικώ πιστεύω ότι η συμβαστική πρόταση πάει προς σωστή κατεύθυνση. Κάποια σημεία βεβαίως πρέπει να τύχουν ε, ε, ε, διευκρίνησης ή βελτίωση και περιμένω να δω την τελική μορφή που θα πάρει η έκθεση της κυρίας Κόμη. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, κύριε Κρόιτσμαν, στην τελευταία έκθεση του κυρίου Κουσνίτς είχαμε φτάσει πιο μακριά, γιατί είχαμε πει να μην συμπεριλάβουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είχαμε κάνει και ακρόαση για να τις συμπεριλάβουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είχαμε τονίσει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα της ε, ψήφου. Ε, δεν θέλω τώρα να μπούμε βέβαια στην, ε, στις λεπτομέρειες, αλλά θα ρωτήσω την Κομισιόν γιατί από τη μία στην, ε, στη δεύτερη εκδοχή λέτε ότι αυτό θα μπορού, ίσως να μην μπορούσε να καλυφθεί από πλευράς κόστους, αλλά στην τρίτη εκδοχή λέτε ότι διατίθενται επιπλέον πόροι. Οπότε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό νομίζω δεν έχει καλυφθεί και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Μιλούμε όμως για εκπροσώπηση, έτσι, μιλούμε για εκπροσώπηση. Και επίσης να πω στην κυρία Κόμη, για την, θα ήθελα να συμπεριλαμβάνουμε στις ακροάσεις όλους τους ε, μπλεκόμενους φορείς, ας πούμε τους ε, εκπροσώπους από, το, από την ΕΚΟΣ. Δεν τους έχουμε συμπεριλάβει αυτούς. Και επίσης τους εκπροσώπους των, συνδικαλιστών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν έχουμε συμπεριλάβει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καλύπτουμε όλους όσους ενδιαφέρονται για την έκθεση αυτή είναι απαραίτητο. Για την Κομισιόν τώρα. Η Κομισιόν νομίζω ότι έχει θέσει τα σωστά ερωτήματα. Ε, θέλω απλώ να θυμίσω ότι για την οδηγία και τα παιχνίδια είχαμε πει ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά τον καθορισμό των ορίων θορύβου. Η Κομισιόν πρέπει να ορίσει συγκεκριμένα όρια ε, χορύπανσης για τα παιχνίδια. και να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο μάλλον λείπει, κατά την άποψή μου. Όλα τα ερωτηματικά, όλα τα θέματα που έχετε θέσει, ναι, απλούστευση, ε, επιτάχυνση, ε, ευελιξία, όλα αυτά είναι καλά. Αλλά η διαφάνεια που είναι. Κάπου πρέπει να μπει και μια πτυχή διαφάνειας. Δεν νομίζω ότι έχει καλυφθεί επαρκώς ε, σχετικά με την εντολή που θα δοθεί για τον καθορισμό των προτύπων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε καλύτερα προς αυτό κατά τα λοιπά, τα θέματα που έχουν τεθεί όντως είναι σωστά. Ένα ακόμη σημείο, τα, τα πρότυπα ICT. Ε, δεν είναι θέμα αυτό μόνο ε, των δημοσίων συμβάσεων, αλλά νομίζω ότι και, άλλοι, ε, και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πρότυπα ICT. Και επίσης θα ήθελα να κάνουμε και μια συζήτηση για το πώς στον τομέα αυτό μπορούμε να αποφύγουμε να μην είμαστε πολύ αργοί γιατί στον, στα πρότυπα, ε, τα πρότυπα αυτά το, σε αυτόν τον τομέα της ε, τεχνολογίας εξαρτώνται πάρα πολύ από την ταχύτητα. Οπότε, ε, ίσως οι βιομηχανίες μας να μην ε, βρίσκονται στον, ε, να μην ακολουθούν τον τόσο γρήγορο ρυθμό των τεχνολογιών. Στην τελευταίο γύρω συζητήσεων που είχαμε κάνει, είχαμε, όταν είχαμε δηλαδή ε, υποβάλει την ε, έκθεση πρωτοβουλία, ήταν σαφέ ότι για τι υπηρεσίε υπάρχει και ανάγκη των, των αγορών. Υπάρχουν οι ανάγκε των αγορών που πρέπει επίση να αναφέρονται. Και εκεί επίση θα πρέπει να γίνει κάτι για την τυποποίηση. Οπότε πρέπει πιο ε, συγκεκριμένα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε και πού θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Well, I think your suggestion about Νομίζω ότι η πρότασή σας για την ένταξη ορισμένων από τις έρωτα της ακροάσεων, της ακροάσεως μάλλον στη συζήτησή μας δεν είναι καθόλου κακή. Ήδη έγινε συγκεκριμένη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα και σε σχέση με τα του ICT και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι σκιώδεις θέλουν να πούνε κάτι. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Θα ήθελα να επανέλθω στην αρχή της συζήτησης, όταν τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τους υπόλοιπους εισηγητές το θέμα ε, για το θέμα το οποίο θέσατε. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε η τυποποίηση και γενικότερα να μην δημιουργήσει μια εξάρτηση επιβαλόμενη μάλιστα εκ των άνω. Από την άλλη επιθυμούμε η τυποποίηση να παραμείνει ένα μέσο ανταγωνιστικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι η έκθεση αυτή και χάρη στην εισηγήτρια και χάρη στην, ε, στους υπόλοιπους συναδέλφους είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε οι περισσότεροι. Αν διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας ε, του αντίστοιχου οργανισμού, αν ενισχυθεί ο ρόλος των αντίστοιχων εθνικών οργανώσεων, Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Άλλωστε έχει ισορρευθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετή εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο είναι περισσότερο τεχνικό θα έλεγα και όχι τόσο πολιτικό. Και η Επιτροπή με την δική της αξιολόγηση των επιπτώσεων δείχνει πως μπορούμε να διευρύνουμε τη συζήτηση αυτή. Να αναφερθώ στο θέμα της ταχύτητας. Ε, όταν εγώ ίδιος ξεκίνησα την έκθεσή μου, ναι, ο κύριος Κότσουσνικ, διαπίστωσα ότι υπήρχαν αρκετές πιέσεις ε, έτσι ώστε οι κανόνες να τεθούν σε ισχύ με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό δεν είναι κακό από μόνο του. Από την άλλη απαιτείται κάποιος χρόνος έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα των προτινόμενων ρυθμίσεων ότι είναι γρήγορο δεν είναι υποχρεωτικά και σωστό, ιδιαίτερα στον τομέα που μας ενδιαφέρει εμάς κάτι τέτοιο σίγουρα δεν είναι σωστό. Πήραμε λοιπόν πάρα πολλές απαντήσεις. Θα τεθεί και το θέμα των δικαιωμάτων ψήφου σχετικά με τη χρηματοδότηση της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, λέει ο Πρόεδρος. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κόμη για να κλείσει τη συζήτηση και να μας παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε τη διαδικασία. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι μια μικρή έκθεση όπως βλέπετε εδώ, έχει πολλές σελίδες. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στην έκθεση αυτή Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που απαντούν στις ερωτήσεις. Και γι' αυτό δίνω τώρα πια το λόγο στην κυρία Κόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά την οποία έκανε. Το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο και σύνθετο. Από την άλλη εμείς έχουμε ανάγκη να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια καλύτερη παρουσίαση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των stakeholders γενικότερα. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα σημεία τα οποία ε, θέσατε, τα υπέρ και τα κατά στα οποία αναφερθήκατε νομίζω παίζουν σημαντικό ρόλο η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες είναι καθοριστική. Αναφερόμεθα σε ένα ιδιωτικό, εθελοντικό, εθνικό σύστημα. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τη διαβούλευση και προς τις ε, stakeholders, σε όλους τους εμπλεκομένους. Θα συνεχίσει λοιπόν η διαβούλευση και βασικός στόχος είναι να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις θέσεις ε, σε χρόνο ο οποίος ε, θα είναι ικανός για να ε, μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά. Για την ταχύτητα εφαρμογής τώρα υπάρχουν διαφορές κατατομής. Ορισμένοι τομείς απαιτούν για λόγους ποιότητας θα έλεγα μεγαλύτερους χρόνους. Σε κάποιους άλλους τομείς μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Μιας και μιλάμε για ένα ιδιωτικό σύστημα, τότε το θέμα του χρόνου θα επιβληθεί από την ίδια την αγορά. Αν έχουμε ένα στάνταρ ας πούμε τριών ετών για ένα τηλέφωνο κινητό κτλ, τότε θα έχει ξεπεραστεί από την αγορά. Πρέπει λοιπόν από τη μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμικές δομές να απλοποιούν την διαδικασία, να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, από την άλλη δεν θα πρέπει να βιαστούμε γιατί αυτό μπορεί να είναι εις βάρος της ποιότητας. Μια μικρή αναφορά τώρα στην ακρόαση. Έχω σταθεί ιδιαίτερα στη συμμετοχή μας σε αυτή την ακρόαση έτσι ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι μία από τις πιο ισχυρές φωνές μπορεί να είναι αυτή η ένωση των επιχειρήσεων η οποία να επηρεάσει και να ορίσει αν θέλετε και τις επιθυμίες του καταναλωτή. Ε, ο στόχος είναι ακριβώς η προστασία του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι, ε, δεν σημαίνει μάλλον ότι δεν θα λάβουμε υπόψη μας άλλες οργανώσεις, αλλά σε συνεργασία με τους υπευθύνους της ΆΝΕΚ ζήτησα να κάνουν μια παρουσίαση 360 μοιρών, να καλύψουν δηλαδή θέματα στα οποία κανονικά αναφέρονται άλλες ενώσεις. Αναφέρομαι εδώ και στο χρονοδιάγραμμα για να μου πείτε αν συμφωνείτε. 23 Νοεμβρίου, ακρόαση. Όχι το απόγευμα, αλλά το πρωί. Προθεσμία για την κατάθεση της πρότασης έκθεσης είναι 22 Δεκεμβρίου. 24 και 25 Ιανουαρίου οι πρώτες συζητήσεις, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 7 Φεβρουαρίου, εξέταση τροπολογιών 28 και 29 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 20 Μαρτίου και νομίζω ότι τον Μάιο του 12 μπορούμε να φτάσουμε στην Ολομέλεια, ενδεικτικά το λέω αυτό. Βλέπετε ότι δεν είναι ένα πάρα πολύ χρονικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, αλλά παρόλα αυτά μας δίδει το χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά, είναι απαραίτητο αυτό, πρόκειται για έναν κανονισμό θυμίζω και όχι απλά μια οδηγία και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε με το χρόνο που χρειαζόμαστε τη σημασία του εγχειρήματο. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους, είμαι απόλυτα διαθέσιμη. Uh, well, thank uh, Ευχαριστώ κυρία Κόμη. Ευχαριστώ τους εισηγήτρια λοιπόν και τους σκιώδεις να πω ότι είμαστε σε επαφή με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τα σχέδια προτεραιότητα στα πλαίσια της ενιαίας πράξης. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε μήπως μπορούμε να μειώσουμε ε, την χρονική διάρκεια αυτού του προγράμματος, αλλά χωρίς να μειώσουμε την ποιότητά του. Αλλά αυτά θα τα αποφασίσει και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Τώρα για το διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν σε διάφορες τέτοιες υπηρεσίες τυποποίησης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που παρακολουθούν την συζήτηση. Αυτό είχε γίνει και με την έκθεση του κ. Κότσουσνικ. Για όλους που μας παρακολουθούν λοιπόν από το διαδίκτυο, τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους. Και στην ιστοσελίδα μας θα υπάρξει μια σελίδα για την τυποποίηση με πάρα πολλούς συνδέσμους σχετικούς με το θέμα κάτι το οποίο θα σας επιτρέψει να παραμείνετε σε επαφή με τα βήματα εξέλιξης και προόδου του συγκεκριμένου θέματος. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό νομοθετικό θέμα, το οποίο αφορά μια πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με, την, με τον σεβασμό και την επιβολή από πλευράς τελωνίων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιούργεν Κρόιτσμαν, εισηγητής. Έχουμε και την κυρία Γκάλο, την κυρία Χέντς, τον κύριο Ένστρομ. Ο κύριος Μακλόκιν δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε αρκετά σημαντική παρουσία σκιωδών. Εγώ σε λίγη ώρα θα πρέπει να φύγω και θα με αντικαταστήσει η συνάδελφος και καλώ τον κύριο Κρόιτσμαν να ξεκινήσει τη συζήτηση σε ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι δίνουν κίνητρα στην έρευνα για την, ε, και, στην ε, επένδυση για την ανάπτυξη. Αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ανθρωπότητας ανεξάρτητα από, την, ε, από το μέγεθος της κάθε χώρας τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν το 81% των, α, ε, ε, ε, της καταγραφής της, από την Standard Poor's. μπορούν να ε, βοηθήσουν στην ε, προφύλαξη της ε, δημόσιας υγείας των καταναλωτών. Μιλούμε κυρίως για πνευματικά δικαιώματα για τα παιχνίδια, για τα ιατρικά προϊόντα, για τα σαμπουάν, για καλλιτικά, για διάφορα. Πρέπει βεβαίως να έχουμε μια καλύτερη συγκριτικά θέση για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα, να εξασφαλίσουμε μάλλον τα πνευματικά δικαιώματα. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε τον κανονισμό 1383 του 2003 της Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα αυτά και να τα προστατεύσουμε, καθώς επίσης και να τα συμπεριλάβουμε στην εσωτερική αγορά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης 2009-2012. Η επέκταση σε πνευματικά δικαιώματα και για, την, και για άλλους δομείς είναι πολύ σημαντική. Το προβληματικό μόνο είναι ότι η εφαρμογή χρειάζεται περισσότερους πόρους, κάτι που αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι δύσκολο να υπάρξει. Κατά 92% προστατεύτηκαν, ε, τα, ε, προστατεύτηκαν οι καταναλωτές το 2010 μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων. Ε, οι τελωνιακές αρχές επίσης ε, έχουν, μπόρεσαν να καταγράψουν πολύ περισσότερες ε, περιπτώσεις κατάχρησης των πνευματικών δικαιωμάτων. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν καλύτερες κατευθυντήρες γραμμές για τις τελωνιακές αρχές. έτσι ώστε να μπορεί η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων να είναι πολύ καλύτερη. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διεκτικών αρχών, των τελωνιακών αρχών πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις παραβάσεις των καταπάτησης ε, ε πνευματικών δικαιωμάτων και σε τρίτες χώρες οι εταιρείε αποστολή θα πρέπει να υποχρεούνται να καταγράφουν τις πληροφορίες και να τις δίνουν, ε, τις, να δίνουν τις πληροφορίες στις αρχές για την ε, προέλευση των ε, φορτίων που μεταφέρουν. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις εταιρείε τέτοιων μεταφορών, οι οποίοι πολλές φορές αποτελούν, κάνουν καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης πρέπει να δούμε εάν ήταν, αν είναι σκόπιμο στις τελωνιακές αρχές να δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουν τους ε, ε αποστολείς, τους, ε, τα στοιχεία, τα, δεδομένα των ε, ε, όσων εμπορεύονται τα πακέτα προς μεταφορά. Μιλούμε για χώρες όπως η Βουλγαρία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Φιλανδία ε, Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει και συγκατάθεση του ιδιοκτήτη να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία εφόσον αυτό δεν ε, έχει, δεν έχει, εφόσον δεν έχει παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού μέσα σε μια συγκεκριμένη ε, χρονική περίοδο. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα την προστασία των α, πνευματικών δικαιωμάτων. Η δυνατότητα αυτά τα εμπορεύματα να καταστρέφονται και αυτό να επαφείται μόνο, ε, σε, μόνο στις ε, αρχές ίσως να είναι ε, πολύ επιβαρυντικό για τις τελωνικές αρχές και σε ό,τι αφορά το κόστος. Από το 2009 μέχρι το 2010 τριπλασιάστηκαν αυτές οι περιπτώσεις Επίση, τα μικρά πακέτα, είναι, οι μικρές αποστολές δεν έχουν οριστεί επαρκώς στο κείμενο, γιατί σε αυτές τις ε, μικρές αποστολές πολλές φορές ε, καταπαντούνται σημαντικά όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Επίση θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο όριο κατόφλι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνούμε. Υπάρχει μια ομάδα ε, θα πρέπει να υπάρξει μάλλον μια ομάδα εργασία από την Κομισιόν η οποία να ελέγξει τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα, τι γίνεται με τη βιομηχανία. Είναι προ όφελο ε, όλων να υπάρξει μια ρύθμιση του τομέα αυτού. Η διευκρίνηση του των ε, κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, η προστασία τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ευθύνη που έχει ο κάτοχος είναι επίσης σημαντική. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το ποιος τελικά καταστρέφει τα ε, προϊόντα τα οποία έχουν ε, μεταφερθεί και με κάποιο τρόπο έχουν καταπατήσει τα, τα πνευματικά δικαιώματα. Θα δημιουργηθούν έτσι τα κίνητρα για τις εταιρείες αποστολής, μεταφορών, και να σας πω και κάποια παραδείγματα. Όταν ας πούμε ο κάτοχος των δικαιωμάτων θέλει να καταστρέψει τα προϊόντα και μετά ε, καταλήγει να είναι αυτός, αυτός που φταίει, προφανώς ε, καταλαβαίνετε ότι έχει υπάρξει πρόβλημα. Ξέρω ότι δεν το ακούτε ευχάριστα αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να υπάρξει υποχρέωση. Αν τελικά δίνουμε ε, προστασία των ε, κατόχων, διότι δεν μπορούμε πρώτα να του δίνουμε ε, το δικαίωμα και μετά να του κατηγορούμε για το ότι θέλουν να καταστρέψουν τα προϊόντα τα οποία έχουν καταπατήσει το δικαίωμα που κατέχουν οι ίδιοι. Βεβαίω αυτό θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και διασυνοριακά, εφόσον υπάρχουν οι εγκαταστάσει και ο κάτοχο μπορεί να αναλάβει το κόστο. Προ το παρόν, στη χώρα όπου γίνεται η καταπάτηση, πρέπει να γίνει και η καταστροφή των προϊόντων. Α πούμε, στο Λουξεμβούργο, που είναι μικρή χώρα. Εκεί όμως δεν υπάρχουν οι ε, ε, κατάλληλες οπότε στις γειτονικές χώρες του Λουξεμβούργου που υπάρχουν εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να γίνουν άνετα οι καταστροφές. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών. Στον ε, κανονισμό επίσης λέει ότι τα προϊόντα που έχουν ε, πνευματικό, που έχουν πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει να αποστέλλονται πίσω εφόσον έχουν καταπατήσει ευρωπαϊκά δικαιώματα παρόλο που μπορεί να προέρχονται από ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Αμερική ή από τρίτες χώρες. Θα πρέπει βεβαίως οι αρχές να αξιολογούν το αίτημα καταπάτησης ε, των ε, δικαιωμάτων Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, εξασφάλιση της ε, πρόσβασης στην, ε, στα διάφορα προϊόντα. Ο κανονισμός όμως δεν διαχωρίζει μεταξύ των γενώσιμων φαρμάκων και των υπόλοιπων φαρμάκων. Μπορεί πολλέ φορέ αυτά τα προϊόντα να περιλαμβάνουν δηλητηριώδει ουσίε ή τοξικέ ουσίε, γιατί μπορεί να είναι ψευδεπίγραφα. Και είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τις διατάξεις για τις ε, περιπτώσεις αυτές. Τα κριτήρια για, θα, για, την, για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν καλύτερα. Θα σταματήσω εδώ και να σας πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Με τους, ε, με τους κοιόδης είπαμε ότι στις 22 ε, θα το ξαναδούμε θα, μεταξύ 15 και 30 του μηνός θα κάνουμε μία ακρόαση για την ε, σωστή εφαρμογή στην, ε, των τελωνιακών αρχών, των ε, προτύπων αυτών που υπάρχουν για τα εγκαταπάτηση των δικαιωμάτων, κυρίως για τα διαμετακομιζόμενα ε, προϊόντα. Οι σκιώδεις την ξέρουν τη συζήτηση αυτή και συμφωνούν. Η Κομισιόν μας ε, ζήτησε να ε, ε, επιταχύνουμε λίγο την όλη διαδικασία, οπότε μετά την ακρόαση, αρχές Δεκέμβρη 2011, θα αποστείλουμε την έκθεση για μετάφραση. Στις 9 Γενάρη θα, έχουμε το σχέδιο, θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε 20 Ιανουαρίου προθεσμία για αποβολή τροπολογιών. Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, μπορούμε να συζητήσουμε τις συμβαστικές πρωτοβουλίες. Μετά έχουμε την ψηφοφορία στις 28 Φεβρουαρίου και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις 28 Μαρτίου. Οπότε από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που ήταν για το Μάη, έχουμε πάει δύο μήνες πριν και γίνεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Μάρτιο, τέλος Μαρτίου. Ελπίζω να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα τη ε, Κομισιόν. Αυτά και ευχαριστώ. Bonjour à toutes et à tous. Καλημέρα σε όλες και όλους. Αναλαμβάνω εγώ την Προεδρία τώρα. Κύριε Κρότσμαν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της εκθεσής σας που ήταν τόσο πλήρης για ένα τόσο σημαντικό θέμα και συγχρόνως περίπλοκο και δύσκολο. Μας ετοιμάσατε ένα κείμενο για την πρώτη συζήτηση πάρα πολύ πλούσιο. Γι' αυτό και θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδες συζητητές με τη σειρά. Η κυρία Γκαγιό πρώτα, μετά μετά ε, ο κύριος ε, Η κυρία Χάρκιν δεν είναι εδώ. Και μετά στον κύριο Ντεγιόγκα. Γιατί ε, ο κύριο Σακίν είναι εδώ. Η Μαριέλ Καγιό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επενθυμίσω κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιεύει 14 2011 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4.000 κατασχέσεις το 2010 από τα τελωνία που είναι το διπλό από τις κατασχέσεις που είχαμε το 2009. Πάνω από 103 εκατομμύρια προϊόντα κατασχέθηκαν. Σας κατακλείσω εδώ με νούμερα, αλλά είναι γιατί πρόκειται για μια πρακτική η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στις θέσεις απασχόλησης βέβαια. Εξάλλου, όπως είπε και ο εισηγητής, Πρόκειται για πρακτική η οποία απειλεί και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θεώρηση του κανονισμού και μια που είμαστε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να περιορίσω τις παρατηρήσεις μου σε τρία σημεία. Πρώτον, εύρος εφαρμογής του κανονισμού. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η έκταση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και από την άλλη μεριά υπάρχει οι περιπτώσεις ε, στις οποίες μπορούν να παρεύουν τα τελωνία. Για το πρώτο στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής να καλύψει όλα αυτά τα θέματα και για τις γεωγραφικές ενδείξεις κλπ. Αλλά από την άλλη, θα ήθελα να ξέρω την άποψη και του συγκητή αλλά και όλων των άλλων συναδέλφων που ενδιαφέρονται για το θέμα, για το κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παράλληλες εισαγωγές. Υπενθυμίζω ότι οι παράλληλες εισαγωγές έχουν να κάνουν με αυθεντικά προϊόντα και ότι οι τελωνιακές αρχές δεν έχουν πάντα στη διάθεσή τους το συμβόλαιο ή την ε, σύμβαση. Άρα είναι δύσκολο για τους τελωνιακούς να ξέρουν κατά πόσο οι συμβατικές υποχρεώσεις τηρούνται ή όχι. Εξάλλου, μαθαίνουμε ότι πολλές παράλληλες εισαγωγές συνυπάρχουν και συνταξιδεύουν με εισαγωγές οι οποίες ε, είναι ψευδεπίγραφα προϊόντα, πλαστά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξέρω, θα συμπεριλάβουμε ή όχι τις παράλληλες εισαγωγές και πώς θα φροντίσουμε ώστε τα τελωνία να έχουν χρήσιμες πληροφορίες για να μπορούν να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Εξάλλου πρόκειται για νέα καθήκοντα, άραγε ε, αποτελεί ήδη καθήκον τους. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να δούμε. Λοιπόν, πάντα σχετικά με το εύρος εφαρμογής και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να παρέμβουν τα τελωνία. Εγώ σημείωσα την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η οποία αποκλεί από το εύρος εφαρμογής του κανονισμού το τράνζιτ φαρμάκων. Γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, έπρεπε να υπάρχει η εξαίρεση αυτή για να μην βρεθούμε σε διαμάχη στον ΠΟΕ. Απ' την άλλη όμως, όταν διαβάζω το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συνειδητοποιούμε ότι τα ψευδεπίγραφα φάρμακα τον Ιανουάριο του 2010 έχουν να κάνουν κυρίως με τις αφρικανικές χώρες, ε, την Ασία, την Λατινική Αμερική, όλες τις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική οικονομία και εκεί είναι που απαντάτε περισσότερο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για αυτή την πραγματικότητα και να καθίσουμε και να σκεφτούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή ή όχι. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι κάτι το οποίο ανέφερε και ο εισηγητή μα και έχει να κάνει με τι ταχυδρομικέ αποστολέ. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι γεγονός ότι τα... η αποστολή με το ταχυδρομείο πλαστών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά πολύ. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει μια ειδική διαδικασία για την καταστροφή εμπορευμάτων όταν πρόκειται για μικρά πακέτα, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να διευκρινίσουμε με ποιο τρόπο θα προχωράει η διαδικασία αυτή έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 διαβάζουμε ότι προβλέπεται μια προθεσμία 20 ημερών. 20 μέρες ώστε αυτός που κατέχει το εμπόρευμα να μπορεί να μεταφέρει την άποψή του. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη η περίοδος αυτή και δεν έχει καμιά σχέση με την περίοδο επαλήθευσης της ε, αλκοολεμίας, για παράδειγμα, του ποσοστού αλκοόλ. 20 μέρες για να μπορεί να εκφραστεί ο κατέχον το εμπόρευμα μου φαίνεται πολύ. Η παράγραφος 7 τώρα λέει ότι η καταστροφή γίνεται υπό τελωνιακό έλεγχο και με έξοδο των τελωνιακών αρχών. Ναι, αλλά σε τι βαθμό εδώ έχουν την ευθύνη οι τελωνιακοί. Αυτό δεν το λέει και αυτό πρέπει λοιπόν να το δούμε. Το τρίτο μου σημείο για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και μετά θα σταματήσω είναι το εξής. Οι διαδικαστικές εγγύσεις είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα να ακουστεί η άποψη αυτού που κατέχει τα προϊόντα, το προϊόν, το εμπόρευμα, γιατί θεωρείται πάντα αθώος, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Η προθεσμία αυτή των 20 ημερών, σας είπα, ότι μου φαίνεται πολύ εξάλλου μπορεί σε αυτή να προσθεθούν και, άλλα, και άλλες καθυστερήσεις. Η τελευταία μου ερώτηση λοιπόν είναι εξή. Ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια που ανακρίνεται ο κατέχων τα εμπορεύματα αυτά. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Να, τρία σημεία που ήθελα να θίξω σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μαριέλ. Θέτεις ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Πράγματι είναι σημαντικό να δουλέψουμε καλά, παράλληλα, αλλά και φροντίζοντας να υπάρχει αρμονία ανάμεσα σε εμά και στην Επιτροπή ΜΚΑ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Άννα. Άννα Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Αυτό που μπορώ να σας πω ευθύ αμέσω είναι ότι βρίσκω πολύ θετικό να μπορούμε να δουλέψουμε με τον εισηγητή πάνω σε αυτά τα θέματα. Οργάνωσε πάρα πολύ καλά το χρονοδιάγραμμα, τις συνεδριάσεις με τους κοιόδες εισηγητές και αυτό είναι πολύ θετικό. Πιστεύω ότι έγινε μια καλή δουλειά. Είναι ένα θέμα που έχουμε ήδη θίξει πολλές φορές μέχρι τώρα. Χρόνια συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Τα συζητήσαμε όταν ήμασταν στην ασφάλεια των παιχνιδιών, όταν επίσης ε, συζητούσαμε για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, όταν συζητούσαμε για τα πλαστά ε, προϊόντα, πλαστές ηλεκτρικές συσκευές κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε την οπτική γωνία του καταναλωτή, γιατί αυτό το θέμα, αυτή η οδηγία έχει να κάνει με τον καταναλωτή. Το σημαντικό είναι πώς θα προστατεύεται ο καταναλωτής, η υγεία του κλπ. Επιμένω, πρέπει να σκεφτόμαστε κατά κύριο λόγο και κατά προτεραιότητα τον καταναλωτή. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα το σημείωσα και περιμένω και εγώ το σεμινάριο που προτείνεται και που πιστεύω ότι το ετοιμάζετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ο κύριος Άμστρομ από τους Πρασίνους έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το εξή. Πλαστά προϊόντα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι παράνομο, πρέπει να είναι παράνομο η εισαγωγή τώρα πειρατικών προϊόντων. DVDs για παράδειγμα, για εμπορικό σκοπό, όντως παράνομο, πολύ σωστά. Υπογραμμίζω ότι ακόμα και εγώ βρίσκω ότι είναι παράνομο, ότι δεν είναι καλό. Αλλά κατόπιν τούτων, ο κανονισμός αυτός είναι προβληματικός γιατί πηγαίνει υπερβολικά μακριά. Γιατί επιτρέπει στα τελωνία να κατάσχουν προϊόντα τα οποία δεν είναι παράνομα αυτά καθ' αυτά και θα σας δώσω παραδείγματα. Πρώτον, οι παράλληλες εισαγωγές είναι νόμιμες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές μέχρι τώρα έχει πει και ότι είναι νόμιμα αλλά και ότι πρέπει να είναι νόμιμα. Μίλησα λοιπόν για τις παράλληλες εισαγωγές. Είναι νόμιμες. Γιατί κατασκευάζονται ε, με τη συνένεση του κατόχου της άδεια και μπαίνουν σε κάποια άλλη αγορά. Προσπαθούν να έχουν υψηλότερη τιμή στην Ευρώπη από ό,τι αλλού, δεν θέλουν ε, να καταστραφεί ο ανταγωνισμός. Εντάξει, καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε να έχουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη, αλλά το Κοινοβούλιο δεν έχει εγκρίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Άρα είναι νόμιμες οι παράλληλες αυτές αγωγές. Ενώ με τον κανονισμό αυτό τα τελωνία μπορούν να κατάσχουν νόμιμα προϊόντα. Και αυτό μου φαίνεται με προβληματικό. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο παράδειγμα γιατί λέω ότι πάει υπερβολικά μακριά η ρύθμιση αυτή. Δεύτερον, παράδειγμα. Πλαστά πειρατικά προϊόντα είναι κακά, πρέπει να είναι παράνομα όταν εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς. Όμως όταν μιλάμε για μικρές ποσότητες, ε, για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική, τότε πρέπει να υπάρχει διάκριση. Γιατί αυτό είναι νόμιμο σε πολλές χώρες μέλη. Θεωρείται παράνομο σε μερικές άλλες, αλλά σε άλλες είναι νόμιμο, αν πάμε σε μια ιστοσελίδα. Και βρούμε ένα ζευγάρι παπούτσια Nike, οτιδήποτε, ως πάντων, σε καλή τιμή. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή θεωρείτε ότι είναι αυθεντικό το προϊόν, οπότε είσαστε θύμα και τότε τα τελωνία θα τιμωρήσουν αυτόν. Το θύμα που τα αγόρασε. Μπορεί να, από την άλλη μεριά, αυτό είναι η δεύτερη περίπτωση, να αντιλαμβάνεται ότι είναι πλαστό το προϊόν. Ωραία, αυτό δεν μας αρέσει. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά σε πολλές χώρες είναι νόμιμο παράλληλα αυτά. Ενώ με τη ρύθμιση αυτή τα τελωνία μπορούν να κατάσχουν πράγματα των καταναλωτών, ακόμα και όταν αυτά είναι νόμιμα. Ε, κάλεβα σωστά αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών μας. Γιατί στο κάτω-κάτω γι' αυτό υπάρχει Επιτροπή μας αυτή, γι' αυτό θέλουμε και ρυθμίσεις και κανονισμούς. Αν δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που τελικά αποτελεί ρουτίνα, τα τελωνία, να κατάσχουν πράγματα τα οποία αγοράζουν μέσω του διαδικτύου οι καταναλωτές, για λόγους τους οποίους δεν μπορεί να καταλάβει ο καταναλωτής, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει, δεν θα διαβάσει εξάλλου και την, τον κανονισμό αυτόν. Αν θέλουμε να κάνουμε ζημιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μεταφορές εμπορικών προϊόντων, ας εγκρίνουμε ένα τέτοιο κανονισμό. Άλλες φορές, άλλες εκθέσεις λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη, ότι θέλουμε οι καταναλωτές να νιώθουν ε, ότι είναι προστατευμένοι όταν αγοράζουν μέσω του διαδικτύου. Αν όμως εγκρίνεται ένα τέτοιο κανονισμό που ο καταναλωτής βλέπει ότι κατάσχονται προϊόντα τα οποία αυτός έχει πληρώσει και δεν θα πάρει ποτέ πίσω τα λεφτά του προφανώς, αν κατασχεθούν, αυτό κάνει ζημιά στις προσπάθειές μας. Αυτά είναι τα κύρια μου σημεία. Εντάξει, υπάρχουν και μερικά άλλα σημεία για τα οποία πιστεύω ότι πάει υπερβολικά μακριά ο κανονισμός αυτός, αλλά αυτά ήθελα να σας πω προς το παρόν. Πρόεδρο. ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεγιόνγκ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι λίγο πολύ και εγώ στην ίδια κατάσταση όπως και η κυρία Χέιντ, δηλαδή ότι θεωρώ ότι είναι ένα τεχνικό θέμα αυτό και ο στόχος του είναι πάρα πολύ καλός, συμφωνώ και εγώ. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καταναλωτής να μπορεί να νιώθει εμπιστοσύνη όταν αγοράζει. Η εφαρμογή όμως τώρα του στόχου μου φαίνεται κάπως ε, ασαφής. Δεν ξέρω, θα έχουμε βέβαια και την ακρόση, αλλά εγώ νομίζω ότι χρειάζονται και άλλες διαβουλεύσεις ε, με ταξιάλων και τους καταναλωτές αλλά και τις υπηρεσίες των τελωνίων. Να δούμε, είναι προετοιμασμένοι. Γιατί η έκθεση αντικτύπου, κατά τη γνώμη μου, δεν μου φαίνεται αρκετά πλήρης. Δεν νομίζω δηλαδή ότι καλύπτει όλα τα σημεία. Με απασχολεί λίγο το θέμα αυτό της καταστροφής των προϊόντων και της διαδικασίας που ακολουθείται για την καταστροφή. Νομίζω ότι μερικά πράγματα πάνε υπερβολικά γρήγορα και ότι δεν είμαστε σίγουροι για το αν πρέπει να γίνουν ή όχι. Στους ορισμούς, για παράδειγμα, πρέπει να σας πω επίσης το ότι γίνεται εξαίρεση για μη εμπορικές ε, συναλλαγές Αυτή η εξαίρεση όμως δεν ορίζεται και στα τελωνία ξέρουμε ότι πολλές φορές γίνονται μεγάλες συζητήσεις για κάτι. Είναι εμπορικό, δεν είναι εμπορικό. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι με τους ορισμούς μας. Γι' αυτό θα ήθελα να προετοιμαστούμε καλύτερα, να μιλήσουμε προηγουμένως με τους καταναλωτές, να δούμε αν είναι ικανοποιημένοι. Έπειτα συμφωνώ και με αυτά που είπε ε, που ακούσαμε για τις παράλληλες εισαγωγές. Έχω πάντως ε, εμπιστοσύνη ότι με τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και με την ακρόαση που θα κάνουμε θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ωραία. Είμαστε στην αρχή μόνο μιας ε, συζήτησης που όπως είπα και στην αρχή είναι δύσκολη και περίπλοκη. Χρειάζονται διευκρινήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει πολλές ερωτήσεις για να απαντήσει, θα τη δώσω το λόγο μετά. Κορέα Κάμπο τώρα έχει το λόγο και αν κάποιο άλλο από του ευρωβουλευτέ θέλει το λόγο να μου το πει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανησυχώ λιγάκι από το ότι Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ε, ομιλητή, δεν ακούγεται το μικρόφωνο του. Δεν αναφέρονται πολλά πράγματα για τα γενώσιμα φάρμακα στην ε, πρόταση αυτή. Το πιο περίπλοκο πάντως θέμα, μάλλον τα πιο σημαντικά, είναι οι παράλληλες εισαγωγές και οι αποστολές με το ταχυδρομείο σε μικρά πακέτα. Για το δεύτερο, η μέθοδος εντοπισμού του πλαστού προϊόντος είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο όταν πρόκειται για μικρά πακέτα που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ πολύ αυτά, είναι πάρα πολλά. Έπειτα γιατί απαιτούν και μια τεχνική ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων πάντως έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια με τις εθνικές αρχές προκειμένου δειγματοληπτικά να γίνεται ανάλυση του περιεχομένου των μικρών αυτών πακέτων. Είναι τρομερά τα αποτελέσματα. Γιατί 30 με 50% μέσα σε κάθε τέτοιο πακέτο που περνάει από τα τελωνία περιέχει κάποια μορφή ψευδεπίγραφου προϊόντος. Η ρύθμιση αυτή ασχολείται με αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Δεύτερον, ό τώρα αρχόμαστε στις παράλληλες εισαγωγές. Για τις παράλληλες εισαγωγές συμφωνώ ότι ε, πλήττουν πολλές φορές την φαρμακοβιομηχανία. Όμως, από την άλλη μεριά, επιτρέπουν να έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα για την παραγωγή ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε δεν με εκπλήσει τόσο πολύ το θέμα αυτό των παράλληλων εισαγωγών. Δεν με ενοχλεί τόσο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οι παράλληλες εισαγωγές αποτελούν και ένα μέσο, έναν τρόπο, ώστε πολλά πλαστά προϊόντα να μπαίνουν γενώσιμα φάρμακα, ή άλλα προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Αυτά τα παραδείγματα ήθελα να σας δώσω για να δείξω και εγώ πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είμαστε στην αρχή μόνο μιας περίπλοκης διαδικασίας. Πρέπει να ασχοληθούμε ίσως με αυτό που έχουμε ήδη κρίνει Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και να δούμε τι γίνεται με ό,τι έχουμε μέχρι τώρα εγκρίνει. Πάντως η βοήθεια του συναδέλφου Κρότσμαν και η εκθεσή του είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Κατ' εξαίρεση θα δώσω το λόγο πρώτα στο Συμβούλιο, τον κύριο Σέντα, εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας να μας πει αν συμμερίζεται, εν πάση περιπτώσει, τις ανησυχίες τις οποίες ε, εξέφρασαν οι βουλευτές. Να μας πει επίσης πού βρίσκεται το Συμβούλιο στην εξέταση του συγκεκριμένου θέματος και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Έντερικ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις ίσως όχι σήμερα αλλά πολλές απαντήσεις ερωτηματικά αρκετά σύνθετα. Κύριο Σέντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι ο κανονισμός αυτός για την εφαρμογή των κανονισμών των τελωνίων σχετικά με την πνευματική διοκτησία έχει μεγάλο θα έλεγα νομοθετικό βάρος. Έχει μεγάλο νομοθετικό βάρος ε, και για τον τομέα των τελωνιακών αλλά γενικότερα και για τον τομέα των καταναλωτών πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε ότι οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο την προστασία του καταναλωτή από την είσοδο επικίνδυνων ε, με διάφορους τρόπους προϊόντων, επικίνδυνων ουσιών και θυμίζω ότι οι ουσίες αυτές ε, μερικές φορές μπορεί να φέσουν και σε κίνδυνο τη ζωή την ίδια των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα σχόλιά σας, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Αυτά ακριβώς είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε και στο Συμβούλιο. Αυτά είναι τα θέματα που συζητάει έτσι και αλλιώ και η ομάδα εργασίας που ασχολείται με τις τελωνιακές υποθέσεις του Συμβουλίου και επίσης προσπαθούμε να εξετάσουμε και τις απλοποιημένες διαδικασίες που, ε, ε, για την καταστροφή των ψευδεπίγραφων προϊόντων τα οποία ε, κατάσχονται. Το θέμα τώρα των προϊόντων τα οποία δηλώνει ο ίδιος ο ταξιδιώτης και του μεγέθους, του όγκου ή της ποσότητας των προϊόντων αυτών. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλείται να κρίνει ο τελωνιακός σύμφωνα με τον κανονισμό. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Πολωνικής Προεδρίας ξεκινήσαμε μια πραγματική συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά, άρθρο προς άρθρο. Είμαστε στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης. Η πρώτη ανάγνωση είχε ξεκινήσει, θυμίζω, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας έγιναν τέσσερις συζητήσεις της ομάδας εργασίας και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών τέθηκε και το θέμα του κανονισμού ανάμεσα σε άλλα. συλλέγουμε τις απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων, δηλαδή των υπευθύνων τελωνιακών αρχών, ο εισηγητής παρουσίασε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι και βεβαίως ότι και η αντίστοιχη προσπάθεια την οποία κάνει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα συνδυαστεί με την δική σας προσπάθεια. Πιστεύουμε να φτάσουμε στην τελική φάση της πρώτης ανάγνωσης τον μήνα Νοέμβριο στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία στις αρχές του επομένου έτους. Στην πρώτη συνάντηση που θα γίνει το επόμενο έτος θα είναι μια έκτακτη συνάντηση η οποία θα σφραγίσει ελπίζω ένα βήμα προς τα εμπρός για όλους τους καταναλωτές και τις τελωνιακές διοικήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι οι διοικήσεις των τελωνίων περιμένουν την ομοθετική αυτή πρόταση για να προστατεύσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ε, τα, τα τελωνία τους, την λειτουργία τους. Νομίζω ότι και η ακρόαση την οποία οργανώνεται είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό που θα προσφέρει πολλά στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Κυρία Μέντερη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους όσους πήρατε μέρος στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσουν και τα τελωνία να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις καταπολέμησης των πλαστών και ψευδεπίγραφων προϊόντων. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν. Ερωτήσεις πολύ σημαντικές στα πλαίσια των συζητήσεων τις οποίες έχουμε ξεκινήσει με όλους τους εμπλεκομένους και στο Συμβούλιο. Είμαστε σε θέση τώρα να σας δώσουμε νομίζω τις απαιτούμενες απαντήσεις για να σας επιτρέψουμε και σας να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Αν ξεκινήσει κανείς βασικά με το πεδίο εφαρμογής ε, των πνευματικών δικαιωμάτων που καλύπτονται από τον υποπρόταση κανονισμό σχετικά με τις παράλληλες εισαγωγέ. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Εμείς στοχεύουμε τις παράνομες παράλληλες εισαγωγέ, δηλαδή τις εισαγωγέ οι οποίες δεν έχουν αδειοδοτηθεί, αδειοδοτηθεί συγγνώμη, από τους κατέχοντες τα πνευματικά δικαιώματα. Αν υπάρχουν παρά με την άδεια του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος, σε αυτή την περίπτωση ισχύει η νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός και αν δεν έχει υπάρξει μια τέτοια διοδότηση. Γιατί κάνουμε τη διευκρίνηση αυτή, γιατί όπως είπε και η κυρία Γκαλό, σήμερα τα τελωνία κατά τη διάρκεια των ελέγχων συναντούν προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά προϊόντα, γνήσια προϊόντα, τα οποία όμως είναι αντικείμενο παράνομης παράλληλης εισαγωγής. Συνεπώς, θα ήταν σωστό για τις τελωνιακές αρχές να έχουν την δυνατότητα παρέμβαση στην περίπτωση όπου τέτοιου είδους προϊόντα συναντώνται. Είναι παράνομες, όπως είπαμε, οι μη νόμιμες αυτού του τύπου εισαγωγές. Εμείς δεν αξιολογούμε, δεν κρίνουμε το τι είναι παράνομο ή νόμιμο. Αυτό το κάνει η νομοθεσία που αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι σε ισχύ. Πρέπει όμως να πούμε ότι τα τελωνία που είναι σε θέση να προστατεύσουν και να ζητήσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα αυτά πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Βέβαια για τις τελωνιακές αρχές είναι αρκετά περίπλοκο να καθορίζουν αν μία παράλληλη εισαγωγή είναι πράγματι νόμιμη ή μη. Εμείς εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων, οι οποίοι θα ήθελαν τα προϊόντα τους να εμποδιστεί η εισαγωγή τους, θα πρέπει να δώσουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προς τις τελωνιακές αρχές έτσι ώστε να είναι σε θέση οι τελωνιακές αρχές να εντοπίσουν και να ανοιχνεύσουν ε, σωστά τα προϊόντα. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, το έχουν κατανοήσει οι οικονομικοί μας εταίροι, όλες οι πληροφορίες οι οποίες βοηθούν την αξιολόγηση ενός προϊόντος πρέπει να είναι στη διάθεση των τελωνιακών αρχών. Οι κάτοχοι, οι λοιπόν των πνευματικών δικαιωμάτων ζητούν από την τελωνιακή αρχή να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους και γι' αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ε, έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα τελωνία έτσι ώστε να προστατευθούν τα προϊόντα. Σχετικά με το τράνζιτ, η διαμετακόμιση και σχετικά με τα γενώσιμα φάρμακα. Όπως είχα εξηγήσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που είχαμε κάνει της μελέτης επιπτώσεων, ό,τι περιλαμβάνεται στην έκθεση αντικατοπτρίζει εν πολύ στην συμφωνία η οποία είχε συναυθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου της ε, Ομοσπονδίας της Ινδίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο κανονισμός αυτός είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, διαδικαστικής φύσεως και δεν δημιουργεί συμπληρωματικό δίκαιο σε σχέση με την προστασία η οποία παρέχεται από την ισχύουσα βασική νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόθεσή μας εδώ είναι να διευκρινίσουμε για τις τελωνιακές αρχές ότι όταν κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου προϊόντων διαμετακόμισης ε, βρίσκουν γενώσιμα φάρμακα, όχι πλαστά, όχι ψευδεπίγραφα, αλλά φάρμακα, τα οποία θα τα χαρακτήριζα κανονικά, έγκυρα. Ακόμα και όταν υπάρχει μια προστασία ε, διπλώματος ευαισθητεχνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον έχουν σαν κατεύθυνση μια τρίτη αγορά, μια τρίτη χώρα, το ότι περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν συνιστά λόγο παρακράτησης των προϊόντων αυτών από τις τελωνιακές αρχές. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε το πέρασμα, τη διαμετακόμιση των προϊόντων αυτών προς τρίτες χώρες. Τώρα, για τα πλαστά φάρμακα. Υπήρξε αναφορά και σε αυτό. Υπάρχει μια νέα οδηγία για τα πλαστά αυτά φάρμακα και εδώ πάλι τα τελωνία έχουν το δικαίωμα να παρακρατούν τα φάρμακα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας. Όπως γνωρίζετε η διανομή των φαρμακευτικών ουσιών στην Ευρώπη ε, πρέπει να γίνει μετά από αδειοδότηση των εμπόρων. Τα τελωνία επαληθεύουν εύκολα λοιπόν αν ένα φάρμακο έχει ή δεν έχει την άδεια. Ξέρετε ότι η οδηγία προβλέπει δυνατότητα στο μέλλον για τα τελωνία να δρουν όταν βρίσκουν τέτοιου είδου ψευδεπίγραφα φάρμακα σε διαμετακόμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς ε, προορισμού εκτό της Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς προβλέπεται να υπάρξουν εφαρμοστικέ διατάξεις οι οποίες στην πρακτική θα δείξουν με ποιο τρόπο αντιδρούν και πρέπει να αντιδράσουν τα τελωνία έτσι ώστε να προλάβουμε τα φάρμακα αυτά να βλάψουν την υγεία των καταναλωτών στις τρίτες χώρες. Σχετικά με το δικαίωμα χορήγησης διευκρινήσεων ή εξηγήσεων, αν θέλετε, αυτό είναι μια βασική αρχή βέβαια του δικαίου. Ο καθένας μπορεί να εκθέτει τις απόψεις του, αυτό είναι τμήμα φυσικά και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κοινοτικού δικαίου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε λοιπόν τον τρόπο εφαρμογής του συγκεκριμένου δικαιώματος όταν σε περιπτώσεις ελέγχου ε, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν το συγκεκριμένο δίκαιο επί τη βάση της εθνικής νομοθεσίας και το δικαίωμα αυτό χορήγησης εξηγήσεων ε, έχουν προθεσμίες ίσως μεγαλύτερες από τις 30 μέρες που προβλέπουμε εμείς. και όχι απλά τρεις μέρες όπου απαιτείται η προθεσμία ε, για τον έλεγχο της ε, γνησιότητας ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Λοιπόν, μιλάμε για προϊόντα τα οποία υφίστανται ελέγχους, είναι προϊόντα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του, υπό την κατοχή τη στιγμή του ελέγχου της τελωνιακής αρχής. Εσείς σαν Επιτροπή γνωρίζετε θα έλεγα τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τις νομικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων. Όταν έχει ένα ύποπτο προϊόν η τελωνιακή αρχή έχει στη διάθεσή της 3-24 ώρα έτσι ώστε να κάνει τις απαιτούμενες ελεγκτικές διαδικασίες για το προϊόν και να έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και έχουν τρει μέρες για να γνωμοδοτήσουν προ την τελωνιακή αρχή. Δημιουργούνται λοιπόν αρκετέ καταστάσεις όπου οι τελωνιακέ αρχές πρέπει να επαληθεύσουν τα προϊόντα και παραμένουν τα προϊόντα αυτά υπό την προσωρινή κατοχή των τελωνίων κατά τη διάρκεια της περίοδου ελέγχου. Σχετικά τώρα με τι ε, μικρέ. Euh, là également, je voudrais rappeler que ce que les douanes font euh, est dans la limite de la légalité σχετικά τώρα με προϊόντα τα οποία εισάγονται παράλληλα σε μικρές ποσότητες, προβλέπουμε ότι ο καταναλωτής ή καλύτερο ο μεταφορέας, αυτός ο οποίος παρουσιάζει το προϊόν στο τελωνίο, έχει δικαίωμα να δώσει εξηγήσει μέσα σε ενα εικοσαήμερο. Στην περίπτωση κατά την οποία αρνηθεί την καταστροφή του προϊόντος, εφαρμόζεται η κανονική διαδικασία και ενημερώνεται ο κάτοχος του δικαιώματος ο οποίος μπορεί να προχωρήσει αν θέλετε δικαστικά. Merci Σας ευχαριστώ. Σας άφησα περισσότερο χρόνο γιατί νομίζω ότι έχει σημασία να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα ήδη από αυτό το στάδιο. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο σύντομα στον κύριο Κρόιτσμαν, ευχόμενη φυσικά καλή τύχη σε μια έκθεση τόσο σημαντική για την αγορά και τον καταναλωτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να κάνω ιδιαίτερα σχόλια. Έχουμε την ε, ακρόαση, θα δούμε τι θα προκύψει από αυτήν. Έχουμε το χρονοδιάγραμμά μας, είναι όντως ε, πολύ φορτωμένο. Το καταφέραμε να ε, το πιέσουμε λίγο, να επιταχύνουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ όλους για τις ε, συμβολές τους, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε σε μια καλή έκθεση. Ε, έναν ε, κανονισμό πάντα μπορούμε να τον βελτιώσουμε δίνοντας νέες ιδέες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εκρεμή θέματα που για, το, για τις μικρές ας αποστολές, τα μικρά πακέτα, ε, για τις ε, για, όταν κάποιος έρχεται από τις διακοπές του πόσα, ε, τι μπορεί να κουβαλήσει μαζί του, για να μην θεωρηθεί ότι κάνει εμπόριο. Τέλος πάντων χρειάζονται καλύτεροι ορισμοί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και, τους, και τις θελονικές αρχές αλλά και τους καταναλωτές. Οπότε καλό θα είναι να συνεργαστούμε έτσι ώστε όλα αυτά να βελτιωθούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κρότσμαν και όλους τους άλλους που πήραν το λόγο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια. Συνεχίζουμε με τα τελωνία πάνω σε ένα άλλο θέμα που είναι ο εξυγχρονισμός των τελωνιακών αρχών. Ο κύριος Ματέο Σαλβίνη που είναι εισηγητής απουσιάζει. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Λορέντσο Φοντάνα για να μας παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Ναι, είναι εδώ αυτός. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Σαλβίνη, ο οποίος έχει στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Όταν επιστρέψει θα κάνει ό,τι μπορεί, θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του έτσι ώστε να προχωρήσει η συζήτηση. Θα προσπαθήσω να αντικαταστήσω ε, με τον καλύτερο ελπίζω δυνατό τρόπο και μου έχει αφήσει αρκετές αναφορές τις οποίες θα σας παρουσιάσω. Μιλάμε για τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών υπηρεσιών. Όλοι γνωρίζουμε την σημασία που έχουν τα τελωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και για την πρόσδοση προστιθέμενης αξίας στην εσωτερική αγορά. Το σύστημα των ηλεκτρονικών τελωνιακών ελέγχων νομίζω είναι ο βασικός στόχος έτσι ώστε για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το τελωνιακό σύστημα θα πρέπει να είναι σύγχρονο, ευαίσθητο σε σχέση με τις απαιτήσει των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει εγγυήσει για την ασφάλεια και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Το κλειδί της επιτυχίας του ολοκληρωμένου τελωνιακού συστήματος είναι η έβρεση αυτής της ισορροπίας. Ο ενημερωμένος τελωνιακός κώδεξ υιοθετήθηκε το 2008 για να απλοποιηθούν οι τελωνιακές διαδικασίες και για να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση των τελωνιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο ανανεωμένος αυτός κώδικας δίνει την δυνατότητα να λειτουργήσουν σωστά οι τελωνιακές αρχές των κρατών μελών. Οι βασικές καινοτομίες είναι κάποιες βασικές αρχές σχετικά με το λεγόμενο ηλεκτρονικό τελωνίο, το ενιαίο, εν πάση περιπτώσει, την, την μοναδική θηρίδα ή μονοαπευθυντική, αν θέλετε, στα ελληνικά θηρίδα, το, αλλιώς το one-stop shop που έχει αρχίσει και λειτουργεί. Αυτό μας έχουν πει ότι ικανοποιεί γενικά τους χρήστες των διαδικασιών αυτών και ε, συζητήθηκε ε, στη συνάντηση για την εσωτερική αγορά τον μήνα Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Ιουνίου του 2013 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία υποτίθεται ε, το λεγόμενο ηλεκτρονικό τελωνίο. Δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει. Η εφαρμογή των τελικών τεχνολογιών οι οποίες ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτής της νέας μορφής τελωνιακής αρχής δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί ένας ενημερωμένος κατά τα άλλα τελωνιακός κώδικας χωρίς τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές τεχνολογίες θα είναι ένα σώμα κενό και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πρακτικά και με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή είναι η σκέψη του εισηγητή και αναφέρεται και στο σημείο 8 της πρότασής του. Αυτό το οποίο θα πρέπει να θεωρήσουμε σαν σίγουρο είναι ότι αν υποστηρίξουμε την αναβολή της εφαρμογής του νέου τελωνιακού κώδικα δεν μπορούμε εμείς απλά να περιοριστούμε στον καθορισμό μιας ημερομηνία στο μέλλον γιατί αυτό σίγουρα δεν θα συνιστά ένα θετικό βήμα. Αντίθετα, εμείς θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε σωστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ψηφίζονται και να αποφασίζονται στόχοι οι οποίοι να είναι πραγματικά επιτεύξιμοι και βοηθούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς το ταχύτερο δυνατόν. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν και στο σημείο 11 του ψηφίσματος, και πέρα από τις δυνατότητες εφαρμογή του ενημερωμένου κώδικα, απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο εισηγητής, έτσι ώστε να υπάρχει σταδιακή εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, ξεκινώντας αρκετά νωρίτερα. Ας προσπαθήσουμε μαζί με τις άλλες πολιτικές ομάδες στην φάση κατάθεσης των τροπολογιών να δούμε αν μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια χρονική αν θέλετε προβολή. Οι τελωνιακές αρχές θεωρούνται σαν εκτελεστές αν θέλετε των τελωνιακών ρυθμίσεων. Μετά από την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων ο ρόλος αυτός έχει μειωθεί και στις, στα εξωτερικά μας σίγουρα βέβαια παραμένει σε ισχύ. Αυτός όμως ο ρόλος είναι ένας, υπάρχει άλλος ένας ο οποίος βελτιώνεται συνέχεια, είναι η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των εισαγόμενων προϊόντων. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πάρα πολλοί κίνδυνοι και όχι μόνο τρομοκρατικού χαρακτήρα, να δούμε τι απειλές για την ασφάλεια των καταναλωτών υπάρχουν τα τελωνία δηλαδή θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν σωστά τα πλαστά, τα ψευδεπίγραφα, την τρομοκρατία και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Τα τελωνία είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος έτσι ώστε μόνο ασφαλή προϊόντα και μόνο αγαθά τα οποία υπακούν σε συγκεκριμένες μορφές τυποποίησης θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν του ελέγχου της αγοράς πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα ελέγξουμε τις τελωνιακές διαδικασίες. Το πρόσφατο ψήφασμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή ΙΝΚΟ που έγινε δεκτό στις 8 Μαρτίου σχετικό με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων και τον έλεγχο της αγοράς. Σέλντερ Μόζε ήταν η συνεισηγήτρια. Συνεπώς λοιπόν η έκθεση Σαβίνη αντιμετωπίζει το θέμα της συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές της τελωνιακές και τις αρχές που ελε... τις ελεγκτικές της αγοράς γενικότερα. Ένα άλλο θέμα ε, αφορά την ανάγκη ε, προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παρανόμως εισαγόμενα προϊόντα συνιστούν απώλεια ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραβιάζουν ε, το νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το παραγωγικό ευρωπαϊκό σύστημα και φυσικά και τους ίδιους τους εργαζομένους τους θίγει άμεσα. Γι' αυτό λοιπόν μας απασχολεί στην Επιτροπή μας ε, το θέμα αυτό μέσω της εκθέσεως Κρόιτσμαν την οποία έχετε ήδη ξεκινήσει συζητώντας. Την έκθεση Σαλβίνη λοιπόν υπογραμμίζεται η σημασία καταπολέμησης των πλαστών προϊόντων. Υπάρχει κι άλλος ένας τομέας σημαντικός θα έλεγα για τα τελωνία. Πολλές φορές τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πάρα, πολύ, πάρα πολλές δυσκολίες για την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους τελωνιακούς ελέγχους από τη μία που διασφαλίζουν τη γρήγορη διακίνηση των προϊόντων αλλά και τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων και το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης του κινδύνου αν θέλετε. Αναφέρεται ο Σαβίνης αυτό στο σημείο 5 τα προϊόντα τα οποία δεν παρουσιάζουν κινδύνους πρέπει να εισάγονται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και οι τελωνιακές αρχές να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε προϊόντα υψηλού κινδύνου που προέρχονται από χώρες οι οποίες παραδοσιακά έχουν την τάση μη σεβασμού των ευρωπαϊκών κανόνων και των παραγωγικών διαδικασιών που αναγνωρίζονται σαν έγκυρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε το ότι οι τελωνιακές αρχές των κρατών μελών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σαν να ανήκαν αν θέλετε σε μία ενιαία διοίκηση να λειτουργούν ικανοποιητικά εφαρμόζοντας τους κοινωνικούς κανόνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εναρμονίσουμε συνολικά τον τρόπο, εργασιών, τον τρόπο εργασίας συγγνώμη, των τελωνιακών αρχών στις διάφορες χώρες. Παρ' όλα αυτά προβλέπεται ένα υψηλό επίπεδο εναρμόνισης ανάμεσα στις 27 διοικήσεις των κρατών μελών αλλά πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε τρία βασικά προαπαιτούμενα. Η αποτελεσματικότητα είναι το πρώτο. Τα σημεία 12 και 13 της έκθεσης εδώ είναι ξεκάθαρα. Πλήρη στήριξη στην αρχή της κεντρικής τελωνιακής αδειοδότησης και της εναρμόνισης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Εδώ η συμμετοχή των κρατών μελών θα πρέπει να είναι πλήρη, συνειδητή και αποτελεσματική. Το πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τεθεί σε ισχύ, μάλλον που τέθηκε σε λειτουργία το 2008 και λήγει στο τέλος του 2013, αφορά ακριβώς αυτές τις εναρμονισμένες διαδικασίες. Προωθεί τις συνεργασίες των τελωνιακών αρχών των κρατών μελών μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ε, πληροφορικών συστημάτων. Αυτή είναι η βάση του προγράμματος. Προβλέπεται επίσης ε, και κάποιες κοινέ δράσεις όπως workshop και, ε, και διαδικασίες κατάρτισης. Είναι σημαντικό να προσπαθήσει κανείς το πρόγραμμα αυτό να το θέσει σε λειτουργία για να περάσουμε και σε μια καλύτερη κατανομή των δαπανών που προβλέπονται για τα προγράμματα αυτά και να περάσουμε σε κάποια φάση και σε πιο φιλόδοξες κοινέ δράσεις. Για τις επιχειρήσεις τώρα. Θέλουμε να δοθεί μεγάλη προσοχή στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες πιέζονται από την ανεπάρκεια της τελωνιακής γραφειοκρατίας. Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι τελωνιακές υπηρεσίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Ξέρουμε και τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν. Υπάρχουν ανεπάρκειες, υπάρχουν καθυστερήσεις. Συνεπώς υπάρχει αύξηση του κόστους για την παραμονή, σαν παράδειγμα, των προϊόντων σε εμπορευματικά κυβότια ε, στις υπό τον έλεγχο των τελωνίων περιοχές. Πρέπει λοιπόν τα τελωνία να μην δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη διαφάνεια. Όπως φάνηκε και στην ακρόαση που κάναμε τον μήνα Ιούνιο, έχει μεγάλη σημασία να κατονίσουμε πως η πιστοποίηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να προσδώσει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις με μικρότερη γραφειοκρατία. Αυτά αναφέρει ο εισηγητής στο 14, 15 και 16. Βασικός στόχος είναι να ορίσουμε τον αδειοδοτημένο οικονομικό λειτουργό ή εμπλεκόμενο αν θέλετε. Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας λοιπόν υπάρχει ένας κάποιος αριθμός σήμερα 495 στη Γαλλία, 200 τόσοι στην Ολλανδία και άλλοι τόσοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ μικρή η αριθμή σε σχέση με τον αριθμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρούν ότι συμφέρει τις επιχειρήσεις, ότι τι συμφέρει να προχωρήσουν στην απόκτηση του συγκεκριμένου χαρακτηρισμού. Στα σημεία λοιπόν 24 και 25, όπου αναφέρεται στα θέματα διαφανείας ο εισηγητής στρέφεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διευκόλυνση της ενημέρωσης ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αναγνωρίζετε ότι σε σχέση με το παρελθόν έχουν σαφώς υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού να βελτιώσουμε τις υπόλοιπες πλευρές, να κυκλοφορούμε τις πληροφορίες που δεν είναι χρήσιμες μόνο για μας, αλλά για το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Η διαφάνεια είναι καθοριστική. Είναι κάτι το οποίο εμείς σαν ομοθέτες θα πρέπει να έχουμε πάντα μπροστά μας. Τώρα, σχετικά με την συνεργασία των τελωνιακών αρχών. Στα συμπεράσματα του λέει ο εισηγητής ότι πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία και ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και τα τελωνία, πρέπει να υπάρχει σωστή ανταλλαγή πληροφοριών και χρηστών πρακτικών έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε την αποτελεσματικότητα και τη βεβαιότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται. Τέλος υπάρχει μια πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη της διοικήσεις τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Υπηρεσία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία σοβούν στις αγορές σήμερα. Νομίζω ότι αυτό θα καλύψει τις ανησυχίες και τις απαιτήσει των επιχειρήσεων και των κρατών μελών. Για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, λέει ο εισηγητής ότι η έκθεση συνδέεται και με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνού Εμπορίου και Διλέγχου Προϋπολογισμών. Θα πρέπει να θυμίσω ότι οι τροπολογίες στο κείμενο θα είναι ε, ε, εφικτό να τις καταθέσετε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Ο Σαβίνη μου είπε ότι θα παρουσιάσει αρκετές τροπολογίες έτσι ώστε να ορίσει καλύτερα κάποια από τα σημαντικά σημεία της έκθεσης σχετικά με κάποιες συμβιβαστικές πιθανόν τροπολογίες ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες προτάθηκε η 3η 15 Νοεμβρίου, 3η μεσημβρινή στο Στρασβούργο. Ο Σαλβίνη θέλει επίσης να ευχαριστήσει την γραμματεία της Επιτροπής η οποία ήταν πάντα διαθέσιμη, αρμόδια και ικανή να βοηθήσει. Merci, Monsieur Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φοντανά μπορούμε να πούμε στον κύριο Σαλβίνη ότι πραγματικά μας τα μεταφέρατε σαν να σας ήταν η ο Ήταν πολύ πλήρης η έκθεσή σας. Ευχαριστούμε. Τώρα, το λόγο έχουν οι σκιώδες εισηγητές. Η κυρία Κορκόλα δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σουάπ θα πάρει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Μετά η κυρία Ράπτη. Ο κύριος Σμιτ. Ο κύριος Κονφά. Η κυρία Δερούλε. Ανταυτού, μάλιστα και ο κύριο Δεγιόν μετά. Ο κύριος Σφάτ, λοιπόν έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ, λέει Ιταλικά ο κύριο Βακ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Σαλβίνη για την τόσο μακρά και ενδιαφέρουσα εισαγωγή του και για τη συνεργασία την τόσο καλή που είχε με την κυρία Κορόλα και με τη γραμματεία τη Επιτροπή. Η κυρία Κορόλα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη συνεργασία που είχατε κύριε Σαλβίνη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να προσθέσω τρία πραγματάκια, αλλά θα το κάνω στα γερμανικά αργότερα. Για την προθεσμία για τον, κωδικό, για τον κώδικα των ε, τελωνίων. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει όντως να, υπάρξουν καλύτερη, να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του MCC. Και αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση από τη δική της ε, πλευρά. Ε, ο, η, το, το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού ε, εμπορευόμενου θα πρέπει να συνάδει με ε, τα όσα υπάρχουν διεθνώς, γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι ε, εμπλεκόμενοι είναι σχετικά λίγοι. Το καθεστώς που δίνεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να είναι να αναγνωρίσιμο σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και... Θα πρέπει βεβαίω να γίνεται αυτό μέσω των επίσημων κανόνων τη ε, αμοιβαία αναγνώριση. Η Κομισιόν θα πρέπει να επιτεχύνει τι διαπραγματεύσει στα πλαίσια της, των διαπραγματεύσεων που έχει με τι ΗΠΑ, όπω είπε και η συνάδελφο πριν λίγο, για να βάλουμε και μια πτυχή ελευθερού εμπορίου στην όλη διαδικασία. Κυρία Πρόεδρε, περνάω στα γερμανικά. Να κάνω και εγώ τρία σχόλια που είναι σημαντικά για μένα τι γίνεται με τις προφορικές δηλώσεις στα τελωνία. Ε, θα πρέπει να το κοιτάξει νομίζω αυτό ε, ο εισηγητής. Γιατί μιλούμε για ε, χίλια περίπου ευρώ. Ε, ποσά δηλαδή τέτοια που μόνο προφορικά δηλώνονται στα τελωνία. Ε, νομίζω ότι για τέτοια ποσά είναι σημαντική αυτή η δυνατότητα. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει και ένα, ε, ένα κάποιο πιστοποιητικό με μια σφραγίδα του τελωνιακού για να μπορούν τα προϊόντα αυτά να φύγουν, να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για τέτοιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, ε, έχουμε, ε, που έχουν μόνο μικρά ποσά ή μικρά φορτία θα πρέπει να τους αφήσουμε τη δυνατότητα για να μην τους επιβαρύνουμε ιδιαίτερα. Τώρα, για, τους μη, για την μη τη μη προτιμησιακή προέλευση η προέλευση ενός ε, προϊόντος είναι σημαντική και θα πρέπει να αναφέρεται κατά πόσο έχει υπάρξει μεταποίηση ή επεξεργασία του ε, προϊόντος αυτού. Επίσης, ε, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε ιδιαίτερο τις διαδικασίες, τις διοικητικές για τις επιχειρήσεις και για την εισαγωγή και για την εξαγωγή των προϊόντων θα πρέπει βεβαίω να γίνεται έλεγχος σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για anti-dumping. Επίσης η κατάργηση του first sale rule για τον μηχανισμό αριθμίσης των τιμών. Αν όντως καταργηθεί και δημιουργηθεί προφανώς α, μια πιο αυξημένη τιμή πια για τα τελωνία, θα υπάρξει μεγαλύτερη επιβάρυνση στην, ε, στην βιομηχανία εισαγωγών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομικά το status quo αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στις ε, πρακτικές των ε, επιχειρήσεων. Και οι ΙΠΑ βεβαίως χρησιμοποιούν τον κανόνα αυτό του First Sale Rule. Και νομίζω κυρία Πρόεδρε ότι γενικώ θα πρέπει να τον διατηρήσουμε. Ε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής με τον εισηγητή και προσβλέπω στην περαιτέρω συνέχισή της. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, με τα τελωνία φαίνεται πως κάτι τρέχει. Την πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε για αυτή την έκθεση είχαμε τον blackout. Ε, τη δεύτερη φορά που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε στο Στρασβούργο δεν υπήρχε χρόνος, ήταν κοντά ε, στα μεσάνυχτα. Την τρίτη φορά που προσπαθούμε να συζητήσουμε για τα τελωνία λείπουν οι εισηγητές. Ε, αισθάνομαι ότι μάλλον πρέπει να φύγω κι εγώ και να στείλω αντικαταστάτη <laughs> για να υπάρχει ε, έτσι ομοιομορφία. Τώρα, ο κύριος Σαλβίνη έκανε μια εξαιρετική δουλειά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Φοντάνα θα του μεταφέρει ε, τις απόψεις όλων μας. Και σκέφτομαι, εκεί που είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε, μήπως πήγε για να ε, εργαστεί λιγάκι για το σημείο 6 και την ομοθεσία, δεν ξέρω. Ε, γυρνώντας θα μας πει, φαντάζομαι. Ε, εγώ δεν θα μπω στο περιεχόμενο, ε, γιατί. Γιατί έχω μια συγκεκριμένη προσέγγιση ε, στην οποία, αν σωστά κατάλαβα, υπάρχει μια γενική συμφωνία. Η προσέγγιση την οποία έχω είναι ότι ε, συμφωνούμε καταρχήν όλοι πως πρέπει να παραταθεί ε, η προθεσμία, να πάμε πέρα από το 2013. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο γιατί βλέποντας τα κράτη-μέλη και βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στα τελωνία βλέπουμε ότι δεν επαρκεί ο χρόνος. Άρα χρειάζεται να δώσουμε χρόνο ώστε και τα ηλεκτρονικά συστήματα να προετοιμαστούν σωστά γιατί πάνω εκεί θα βασιστούμε αλλά και οι εθνικοί φορείς να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μου δεν μπαίνω στο περιεχόμενο του κανονισμού γιατί θεωρώ ότι αν μπούμε στο περιεχόμενο ανοίγουμε ε, πολύ μεγάλο πεδίο συζήτησης που δεν θα μας βοηθήσει ε, στην πράξη. Απ' την άλλη πλευρά η έκθεση Κρόιτσμαν που προηγήθηκε και που την ε, βλέπω με πάρα πάρα πολύ καλή διάθεση αγγίζει θέματα περιεχομένου. Και ίσως είναι και πάρα πολύ σωστό εκ μέρους της Γραμματείας και του Προέδρου που μπήκαν και με αυτή τη σειρά να συζητηθούν οι εκθέσεις. Γιατί πραγματικά φαίνεται πόση σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στα ζητήματα. Μένω λοιπόν εγώ στο θέμα της παράτασης και της ανάγκης ε, της παράτασης για την ανάγκη της καλύτερης δυνατής, του καλύτερου δυνατού εξυγχρονισμού ε, των τελωνίων και ε, κάνω μερικές επισημάνσεις για τις οποίες ξέρω ότι ε, εφόσον λείπει ο κύριος Σαλβίνη δεν μπορώ να έχω άμεση απάντηση αλλά θέτω τον προβληματισμό στο τραπέζι για να το δούμε και να δούμε και στις ε, τροπολογίες τι μπορούμε να κάνουμε. το πρώτο ζήτημα είναι η παράγραφος 2 που ε, από ό,τι βλέπω λέει μεταξύ άλλων ε, ο εισηγητής στην έκθεσή του ότι η αποστολή και η εικόνα των τελωνίων πρέπει να οριστούν εκ νέου και καλεί μάλιστα την Επιτροπή να αναδιοργανώσει τη στρατηγική της για τα τελωνία. Εδώ θα ήθελα να έχω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες πώς ακριβώς το σκέπτεται, γιατί μέσα από αυτήν την παράγραφο μπαίνουμε ε, στο περιεχόμενο του κανονισμού και θα ήθελα λιγάκι ε, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες ιδέες. Ε, πάμε στην παράγραφο 13, κεντρικός εκτελονισμός. Ε, τον υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Ε, βάζω όμως έναν αστερίσκο και λέω ότι εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της Κομισιόν. Να έχει τα μάτια της ανοιχτά να υπάρχει συντονισμός και να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής. Ε, κυρίως δε στο σημείο της παροχής πληροφοριών χωρίς εμπόδια ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πάω στο 15 και 16 στις παραγράφους αυτές που αφορούν τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Ε, πολύ σωστά ο κύριος Αλβίνη στην έκθεσή του σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνει κάτι ώστε να μπορούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να έχουν μια παρουσία. Πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν οξυγόνο. Ξέρουμε όλοι, το λέμε συνέχεια σε αυτή την Επιτροπή και πολύ καλά κάνουμε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης. Άρα πρέπει να είμαστε κοντά τους και να μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Ε, συμφωνώ λοιπόν με αυτή την προσέγγιση. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια, ε, στην παράγραφο 15 γίνεται αναφορά σε επιπρόσθετα πλεονεκτήματα για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Και εδώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτά ε, ή πώς το φαντάζεται ο εισηγητής, ώστε να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει καλύτερα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα στο οποίο ε, θέλω να καταθέσω ένα προβληματισμό. Γίνεται αναφορά στο τέλος της έκθεσης σχετικά με τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τελωνίων. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν λάβουμε υπόψη την ανάγκη που έχουμε η Επιτροπή να έχει ένα μάτι, μια φροντίδα, μια μέρημνα για το θέμα των τελωνίων, ίσως θα είχαμε ανάγκη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τελωνίων. Όμως θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Γιατί, Γιατί βλέπω ότι πάμε σε μία ε, πραγματικότητα που δημιουργούμε διάφορες υπηρεσίες σε, στο επίπεδο της Κομισιόν, υπηρεσία για το ένα, υπηρεσία για το άλλο και, και πάει λέγοντας, αλλά στο τέλος ε, φτιάχνουμε υπηρεσίες, έχουμε προσωπικό, αυξάνουμε το οικονομικό κόστος των διοικητικών υπηρεσιών, έχουμε τη σχετική γραφειοκρατία και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ μικρό. Γι' αυτό εκφράζω προβληματισμό σε σχέση με το κατά πόσον είναι ανεγκαία η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τελωνίων. Κλείνοντας, ε, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σαλδίνη και επιφυλάσσομαι για κάποιες τροπολογίες και βεβαίως είμαι ανοιχτή σε συνεργασία. Είσαι πολύ άδικη, Προεδρίνα Μπερναντέτ, πολύ άδικη. Είμαι η μόνη εισηγήτρια που βρίσκομαι εδώ παρούσα και νομίζω ότι μιλάω το λιγότερο δυνατό χρόνο. Ε, ο πρόεδρος έδωσε την εντολή. Τότε είμαι άτυχη διπλά, διότι ήρθε ο πρόεδρος την ώρα που μιλάω. Λοιπόν, κλείνω και λέω ότι επιφυλάσσομαι για τροπολογίες και είμαι ανοιχτή σε συνεργασία βεβαίως και με τον κύριο Σαλβίνη και με τους υπόλοιπους και όδης Ε, Κύριε Πρόεδρε, ε, καλό είναι φαίνεται να μιλάω όταν λείπετε. Έχω συγκριτικό πλεονέκτημα. Καλώς ήρθατε πάντως. Ευχαριστώ, λυπάμαι. Αλλά είναι επειδή περνάει ο χρόνος. Υπάρχουν όμως και άλλοι σκιώδες εισηγητές που είναι στην αίθουσα. Δεν είσαστε μόνο εσείς. Ο κύριος Σμιτ που είναι σκιώδη εισηγητής για τους φιλελεύθερους και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε η οποία αντικαθιστά τον κύριο Κονφάν και στον κύριο Τεγιόνγκ, που είναι σκιώδης εισηγητής και αυτός και στον κύριο Χάρμπερ που είναι επίσης σκιώδης εισηγητής και είναι εδώ. Ε, ε να ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν είδα τους άλλους και όδης εισηγητές. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. That I didn't understand. Ε, thank you and thank you to you, Mr. Fontana. And... Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Φαντάνα. Προσπαθώ να είμαι σύντομος γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση αυτή και ελπίζω η δουλειά που προτείνουμε όντως να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Συζητήσαμε και το χρονοδιάγραμμα και εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν μου αρέσουν οι αναβολές. Το έχω ακούσει πολλές φορές εδώ σε αυτό το σώμα αναβολή-αναβολή και τώρα 2013 δεν είναι αρκετά καλό. Ελπίζω, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με μια άλλη ημερομηνία στόχο, γιατί είναι χρήσιμο. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρνουμε τελικά. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια σημαντική έκθεση αυτή για το ελεύθερο εμπόριο, για την ελεύθερη αγορά και για τα ανοιχτά σύνορα. Είναι εφικτό. Πρέπει να γίνει και αποτελεσματική ρυθμισή αυτή για πολλούς λόγους. Για μένα το κύριο είναι η προστασία της ελεύθερης αγοράς. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό ζούμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Υπάρχουν κάποια ευαίσθητα θέματα εδώ. Κατά σύμπτωση, ο κύριος Σβάμπ αναφέρθηκε σε αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί να ενδιαφέρει τους Γερμανούς πιο πολύ, ξέρω εγώ. Και ο κύριος ε, Κρότσμαν μου τα είπε εμένα. Γίνεται συζήτηση για το όριο των χιλίων ευρώ. Να, βλέπετε, είναι γερμανικό το θέμα. Θα πρέπει να είναι. Γι' αυτό. Άμα είναι γερμανικό, τότε είναι και ευρωπαϊκό. Και υπάρχει και ένα θέμα της προέλευσης των αγαθών, το είπε και ο κύριος Σφαπ. Πρέπει να πω ότι Έχω κάποιες αμφιβολίες για όλες αυτές τις ανησυχίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα θα συμπεριληφθούν στις τροπολογίες μας. Πάντως, για τον κύριο Φοντάνα θέλω να πω τέλος ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι στην ε, έκθεση του κύριου Σαλβίνη, καλώς. Πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτό το σημείο, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ζωτική σημασίας κύρια Πρόεδρε, θα υποβάλουμε τροπολογίες και ελπίζω ο Μάρκο να έχεις μια καλή διάσκεψη. Είμαστε πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς ήρθες πίσω. Bien sûr. Merci pour... Καλώς. Ε, ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Κυρία Ρούλε, θέλετε κι εσείς. Σύντομα. Ένα σχόλιο για το ερώτημά σας. Αν είναι ευρωπαϊκό θέμα ή αν είναι γερμανικό πρόβλημα. Καταρχάς είναι πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κατόφλια. Είναι πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, δεν είναι μόνο γερμανικό πρόβλημα, γιατί εγώ έχω έρθει σε επαφή με πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και ίσω θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Να μην λέμε απλώ ότι είναι γερμανικό πρόβλημα και τέρμα. Είναι πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι μου είπαν, αυτό σα λέω. Εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, υποστηρίζω την πρότασή του, την έκθεσή του. Θεωρώ ότι σε πολλά σημεία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ένα σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω. Κατανοώ τις ε, ανησυχίες του κυρίου Σμιτ και τις ε, ενστερνίζομαι. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε κάτι και να πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν φαίνεται μέσα στην ε, έκθεση και νομίζω ότι θα πρέπει να το συμπληρώσουμε. Γιατί πέραν των, για τη λιτότητα και των πιέσεων των κρατών μελών, νομίζω ότι θα πρέπει να αναδιανεμηθούν οι πόροι και σε ό,τι αφορά το, το, τις ε, τεχνολογίες και τα προϊόντα τεχνολογίας στα τελωνία που πάλι θα έχουν λιγότερους πόρους. Οπότε καλό θα ήταν να ενισχύσουμε την πίεση στα κράτη-μέλη, να το πούμε δηλαδή σαφώς μέσα στην πρόταση, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προχωρήσουν πιο θαραλέα, πιο δυναμικά. Και ένα τελευταίο σημείο, το σημείο 22, έχω μια έτσι, αμφιβολία λέει ότι ε, χαιρετίζουμε την υποβολή της πρότασης από την Κομισιόν. Σήμερα φαίνεται ότι ε, δεν έχει συζητηθεί επαρκώ πια η πρόταση αυτή τη Κομισιόν. σω να πρέπει να είναι λίγο πιο ουδέτερη η διατύπωσή μα στο σημείο αυτό. Πώ να χαιρετήσουμε κάτι που δεν έχουμε συζητήσει καν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεγιόγκ έχει τώρα το λόγο και μετά ο κύριο Άρμπορ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Πιστεύω ότι μας δίνει μια πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε παρετέρω. Τώρα κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για την προθεσμία όπως και άλλοι. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα πετύχουμε ή θα πάει αργότερα για το 2015. Πάντως το βέβαιο είναι ότι το σύστημα όσο προχωράει δεν ε, θα πρέπει να δημιουργούνται εμπόδια εξαιτία καθυστερήσεων σε άλλα σημεία της Ευρώπης, εκεί όπου μπορεί να προχωρήσει δηλαδή. Συμφωνώ με τις δύο παρατηρήσεις του κυρίου Σβάπ πάντως για το όριο των χιλίων ευρώ και για τις ε, ασάφειες όπου εξακολουθούν να υπάρχουν. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πράγματα τόσο περίπλοκα που τελικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως θα θέλαμε. Το επόμενο σημείο μου έχει να κάνει για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Εντάξει αυτά που λέει η έκθεση, αλλά αυτά που δεν λέει είναι πώς θα ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα καλύψουν το κόστος της διαδικασίας αυτής που είναι μεγάλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, ένα σημείο που νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω είμαι ότι είμαι κατά της δημιουργίας μιας νέας υπηρεσίας. Είμαι εντελώ κατά. Εγώ νομίζω ότι για μας ε, είναι περιττό. Δεν μπορώ να τεθώ υπέρ της δημιουργίας μιας νέας τέτοιας υπηρεσίας. Ωραία, σωστό. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ, ο πρόεδρος, που θα έχει και τον τελευταίο λόγο. Ε, πρόεδρος, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όντως σύντομος. Είναι μια εξαίρετη βάση για να προχωρήσουμε, πιστεύω κι εγώ. Ε, έχει το σωστό, τη σωστή απόχρωση και νομίζω ότι πρέπει σε αυτό να βασιστούμε. Τώρα, το θέμα του εναρμονισμένου τελωνιακού κώδικα είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Δεν κρίνουμε τη διαδικασία, πάντως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονός ότι η Επιτροπή αναθεωρεί και χρησιμοποιεί διάφορα νομικά μέσα για να εξετάσει το θέμα είναι καλό. Σίγουρα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τη δουλειά που κάνει. Δεν πρέπει να προχωράμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τα προβλήματα όμω που τίθεται και το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή δεν ελέγχει τελικά όλες τις διευκολύνσεις, όλους τους πόρους. Είναι θέμα κινήτρων περισσότερο. Όμως είναι σαφές ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί ο κόσμο τα περιμένει, τα θέλει πρέπει να καθορίσουμε συστήματα στα οποία να μπορούν να ανταποκρίνονται τα ταλωνία 27 διαφορετικών χωρών. Πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντως στον κόσμο ότι όπως και αν μεταφέρονται τα εμπορεύματα, μην ξεχνάμε ότι οι τελωνιακοί συνήθως κάθονται πίσω από ένα κομπιούτερ και ηλεκτρονικά γίνονται περισσότερες διαδικασίες. Άρα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές για να μπορούν διαφορετικά τελωνίες σε διαφορετικές χώρες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους έγγραφα, πληροφορίες κλπ. Πολλές φορές δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες των τελωνίων ε, πραγματικά. Πολλά από τα εμπορεύματα περνάνε μόνο ηλεκτρονικά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλο και περισσότερες ευθύνες και όλο περισσότερα πράγματα περιμένουμε από τα τελωνία. Εκτός από το θέμα της ασφάλειας, ε, της αντιμετώπισης των πλαστών προϊόντων κλπ. Όμως έχουν τα τελωνία και τα μέσα για να φέρουν σε πέρα αυτά τα καθήκοντα που εμείς τους προσθέτουμε. Λέμε ναι τελωνία, αλλά τα τελωνία δεν προστατεύουν μόνο τα οικονομικά μας συμφέροντα, μέσω δασμών κλπ. Τους ζητάμε να μας προστατεύσουν και από άλλα πράγματα. Τους αναθέτουμε και άλλες ευθύνες που έχουν να κάνουν με τις δικές μας πολιτικές. Πρέπει να έχουν και τους κατάλληλους πόρους λοιπόν, τα μέσα. Τέλος, κάτι άλλο. Το θέμα της νέας υπηρεσίας, όπως είπατε και εσείς, μα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρωί, όταν μιλούσαμε για την τυποποίηση, απέριψε την ιδέα για μια νέα υπηρεσία. Οι ιδέε όμως που αναφέρονται για τη συνεργασία βρίσκω ότι είναι καλές, ιδιαίτερη η ανταλλαγή πληροφοριών. Και έρχομαι και πάλι εδώ στο θέμα των πλαστών προϊόντων και την ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά συστήματα αναφορά, να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίε μεταξύ μα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό για τα τελωνία. Γιατί με τον τεράστιο όγκο προϊόντων που μεταφέρονται, ε, Πώς θα σταματήσουμε ένα πλαστό προϊόν. Πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Συνήθως έρχεται ένα μηνυματάκι και έτσι προχωράμε στην κατάσχεση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μυροσβλίνσκι έχει τώρα το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα έχει το τόσο δύσκολο καθήκον να μας πει την άποψή του πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει χρόνος σχεδόν καθόλου, γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα θέματα τα οποία ετέθησαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε κάποια βασικά θέματα. Όλες οι ιδέες οι οποίες ακούστηκαν θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες από αυτές τις έχουμε ήδη υπόψη μας και είχαμε ήδη στο παρελθόν κάποιες διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πράγματι εμείς περιμένουμε με προσδοκίες πολλές ε, τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναδιατύπωση, αν θέλετε, του τελωνιακού κώδικα δεν μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε εμείς μια νέα συζήτηση γιατί αυτό θα χρειαστεί πολύ περισσότερο κόσμο, χρόνο συγγνώμη, ε, από ότι μέχρι το 2013. Όμως υπάρχει η δυνατότητα, έχουμε ήδη ξεκινήσει και προχωράμε, αυτό είναι στα πλαίσια της κουζίνας της Κομισιόν της Εσωτερικής, ξεκινήσαμε μια διυπηρεσιακή συζήτηση για την αναδιατύπωση του ε, ανανεωμένου τελωνιακού κώδικα. Και θα περάσουμε και σε ένα δεύτερο φόρουμ πριν έλθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις, ε, In για τις Βέβαια το θέμα του χρονισμού είναι κάτι το σημαντικό για μας. Ξέρετε ότι υπάρχει οικονομική κρίση σε, στα κράτη-μέλη, στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη και σε όλα τα κράτη-μέλη η διοίκηση των τελωνίων αντιμετωπίζει προβλήματα περικοπών, οικονομικής συρρήκνωσης κτλ. το θέμα των πόρων των τελωνίων και της αντιστήχησης των πόρων με τις νέες ανάγκες είναι κάτι το βασικό. Για, για το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα υπάρξει μια μαγική ημερομηνία πέρα από την οποία θα έχουν, εφαρμοστούν τα πάντα, θα έχουν εφαρμοστεί τα πάντα. Ο εξυγχρονισμός των τελωνίων και ο εξυγχρονισμός των συστημάτων πληροφορικής είναι διαδικασίες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το ταχύτερο δυνατόν προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας χωρίς να ξεχνάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τώρα για την κυκλοφορία της πληροφόρησης. Εμείς έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, έχουμε δημιουργήσει τα δίκτυα, της ομάδες επαφής και ένα τελευταίο σημείο, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τελωνιακής Υπηρεσίας. Δύσκολο. Ξέρουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε τις εξωτερικές υπηρεσίε. Δεν περιμένουμε ένα θαύμα εμείς εδώ, απλά προσπαθούμε να συνδυάσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις στα συστήματα πληροφορικής έτσι ώστε να επωφεληθούμε όσο περισσότερο γίνεται και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Κατανοούμε τις δυσκολίες που έχουν τα κράτη-μέλη, που ίσως δυσκολεύονται να συνεργαστούν επίσημα, αν θέλετε, σε ένα μαγαζί με πρόσωψη, αλλά είναι αλήθεια ότι λίγο πιο πίσω έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις, απλά δεν έχουν φανεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην επόμενη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φοντάνα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Ευχαριστώ την επιμελητία. Θα μεταφέρετε στον κύριο Σαλβίνη ότι ακούστηκε εδώ. Ο διάλογος που είχαμε ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Υπάρχουν κάποια σημεία διαφωνίας, αλλά υπάρχουν και κάποια κοινά σημεία και θα επανέλθουμε στο θέμα της συζήτησης στην επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ.